Λοιπόν, θα αρχίσουμε αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ξεκινήσω με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης και θα συνεχίσω στην Ιταλική γλώσσα. Το πρώτο λοιπόν θέμα στην ημερήσια διάταξη, η έγκριση της ε, ημερήσια διάταξης. Τα πιο σημαντικά σημεία σήμερα. είναι η παρουσίαση της ειδική έκθεσης της ε, <clears throat> διαμεσολαβήτριας για το Frontex. Προβλέπεται επίσης και η παρουσία μιας αντιπροσωπείας της Επιτροπής Αναφορών του Ιρλανδικού Κοινοβουλίου. Θα ασχοληθούμε επίσης με την υποτιθέμενη διάκριση εις βάρος των λεκτόρων ξένων γλωσσών στα Ιταλικά Πανεπιστήμια. Έχουμε το θέμα της Ισπανίας για την προστασία του περιβάλλοντος στην Αλμέρια και θα αναφερθούμε επίσης και στις επισκέψεις που έγιναν στην Γαλλικία και την Ελλάδα. Θα ασχοληθούμε και με τα θέματα που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων στη Γαλλία και στην Ιταλία. Και τέλος θα συζητήσουμε την έκθεση του 2013 για την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη, η Ευρωπαϊκή Υπηκότητα. Λοιπόν, για κάποια από τα θέματα αυτά θα είναι παρόντες ή υπογράφοντες των αναφορών των σημείων 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12, 17, 18 και 19. Εάν δεν υπάρχουν ε, λοιπόν αντιρρήσεις στην ημερήσια διάταξη όπως πολύ συνοπτικά σας την παρουσίασα, η κυρία Ντάνοσκα έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχω μία μικρή αντίρρηση συμπερίληψη ενό θέματος στην ημερήσια διάταξη και προτείνω να αφαιρεθεί το 16 για την αποστολή στη Γαλλικία, την ερευνητική αποστολή στην Γαλλικία και την εξέταση του εγγράφου εργασίας. Το έγγραφο εργασίας το οποίο λάβαμε για την εξέταση αυτή Έχει ημερομηνία την 28η Οκτωβρίου του 2013 και παρουσιάστηκε μέσω μιας επιστολής που έστειλε η Γραμματεία. Στα πλαίσια αυτής της επιστολής λέγεται ότι αυτή η τελική διατύπωση την οποία προετοιμάσατε και εσείς Πρόεδρε είναι μια συνθετική παρουσίαση όλων των απόψεων των μελών της αντιπροσωπείας στο κομμάτι το περιγραφικό. Εγώ εξέτασα το περιγραφικό κομμάτι και δεν συμφωνώ ότι πρόκειται για μια σύνθεση. Δεν είναι διόλου συνθετικό το κείμενο. Όπως μας εξέγησε και η νομική υπηρεσία, εφόσον υπάρχουν διαφορετικές απόψεις στα πλαίσια του περιγραφικού τμήματος της έκθεσης, θα πρέπει να παρατεθούν και οι διαφορετικές απόψεις. Και στα πλαίσια της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου υπάρχει μια καταπλειοψηφία απόφαση και υπάρχει επίσης και το κείμενο το οποίο ακολουθεί και υπόκειται ε, της διαφορετικής άποψης, της μειοψηφούσης απόψεως. Εδώ έχουμε το αντίθετο. Uh, Εδώ έχουμε ένα ανακάτεμα από δύο έγγραφα. Το ένα έγγραφο αφορά την πλειοψηφία, δύο μέλη, την κυρία Βέρτμαν και την κυρία Σντάνοβκα. Και έχουμε και το κείμενο το οποίο πρότεινε η, ο υπεύθυνος της αντιπροσωπείας, ο Φιλίπ Μπουλάν. Οι δηλώσεις αυτές όμως του κυρίου Μπολάν δεν τίθεται σε εισαγωγικά θα έλεγα. Και αυτό δημιουργεί παρανοήσεις. Ιδιαίτερα για αυτούς οι οποίοι ε, δεν γνωρίζουν το πώς λειτουργεί το σύστημα. Και αν διαβάσει κανείς το κείμενο όσο έχει, μέτρησα ότι υπάρχουν 35 αναφορές του ονόματος του κυρίου Μπολάν και των απόψεών του. Ενώ η δική μας άποψη αναφέρεται έξι φορές. Καλό θα είναι και οι απόψεις των μελών να φαίνονται. Και μερικές φορές λέει κάποια μέλη λέγουν αυτό, κάποια άλλα μέλη λέγουν αυτό. Ποια είναι αυτά τα μέλη, ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά μέλη τα οποία πήγαν ή ενδιαφέρονται για τα θέματα, υπάρχουν και πέντε Ισπανοί μέλη. Σε ποιους αναφέρεται, εν πάση περιπτώσει, η παρουσίαση της επισκέψεως αυτές. Γιατί να παραμένουν ανώνυμα τα μέλη της αντιπροσωπείας και να υποθέτουμε το ποιοι μπορεί να είναι. Δεν πρόκειται λοιπόν για μια ουσιαστική περιγραφή. Πρόκειται για μια ανάμιξη δύο εγγράφων, χωρίς εισαγωγικά, χωρίς αναφορές, χωρίς παύλες. Κάποιες θέσεις που περιλαμβάνονται στη δική μας γνωμοδότηση εξαφανίστηκαν πάρα πολύ απλά και δεν γίνεται καμία αναφορά. Υπήρξε αλλαγή της διατύπωσης. Εμείς εκεί που λέμε υπάρχει σήμερα, αυτό μεταφράζεται υπήρχε κάποτε, χωρίς να υπάρχει εξήγηση γι' αυτό. Συνεπώς λοιπόν αυτό δεν είναι το τελικό έγγραφο εργασίας ε, το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί από την Επιτροπή και προτείνω παρακαλώ να διαγραφεί το άρθρο 10, η έκθεση του άρθρου 16 και να δούμε τι θα κάνουμε από εκεί και πέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα υποστηρίξω τη συναδέλφωσή ήμουν και εγώ μέλλον της αντιπροσωπείας αυτής και καλό θα είναι να πάρουμε το έγγραφο της ε, Τατιάνα και να πάρουμε και την ε, έκθεση του κυρίου Μπουλό και να τα συνδυάσουμε. Γιατί εκεί που λέμε ότι ο κύριος Μπουλάν λέει αυτό, θα πρέπει να πούμε ότι και ο κύριος Μπουλάν λέει το άλλο. Υπάρχουν σημεία στα οποία αναφέρονται οι τοπικές αρχές, σαν παράδειγμα, στη δική μας ε, έκθεση. Και αυτές οι δηλώσεις των τοπικών αρχών στο κείμενο το οποίο μας προτείνεται εξαφανίστηκαν. Ενώ ένα τέτοιο έγγραφο θα πρέπει να αντικατοπτρίζει αυτά τα οποία έγιναν, αυτά τα οποία είδαμε και αυτά τα οποία ακούσαμε. Αυτό δεν σημαίνει ε, ότι ε, θα πρέπει να γίνονται τέτοιου είδους αυθαίρετες παρουσιάσεις. Κοιτάξτε, ακούσαμε και την άποψη της νομικής υπηρεσίας. Γνωρίζουμε ποια είναι η διαδικασία και αυτό το οποίο έγινε είναι απαράδεκτο. Ε, δεν μπορεί κάποιος να αποφασίσει με διαφορετικό τρόπο. Πρέπει να ακολουθηθούν οι σωστοί κανόνες. Αλλιώς αν δεν προστατευόμεθα από τους ίδιους τους κανόνες ε, δεν μένει τίποτα πια. Πρέπει να γίνει μια πραγματική έκθεση η οποία να εξεταστεί στην επόμενη συνάντησή μας, ο κ. Κάσμαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ συμφωνώ με την πρόταση της κυρίας Ντάνοκα να αποσυρθεί παρακαλώ από την ημερήσια διάταξη έτσι ώστε όλες οι πλευρές να μπορέσουν να συναντηθούν και να παράγουν μια έκθεση η οποία να τύχει τη συμφωνία των υπολείπων. Γιατί πρέπει πράγματι αυτές οι εκθέσεις να αντικατοπτρίζουν το τι έγινε, το τι υπόθηκε και το τι είδαμε όταν πήγαμε εκεί. Ε, ευχαριστώ ε, που μου δώσατε το λόγο. Θα πρέπει να δούμε πώς παρουσιάζεται η κατάσταση, γιατί είναι αλήθεια ότι τα μέλη της αντιπροσωπείας που πήγαν στην συγκεκριμένη αποστολή μπόρεσαν να συνεισφέρουν στο περιεχόμενο της συγκεκριμένης έκθεσης. Δεν πρέπει να υπάρξει αναβολή νομίζω. Γιατί αν το αναβάλουμε τότε φοβάμαι ότι αυτή η αναβολή μπορεί να συνεχιστεί επαόριστον. Και αυτό μόνο και μόνο γιατί τελικά να μην ξεχνάμε ποιο είναι το πρόβλημα, ότι δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν μεταξύ τους οι συμμετέχοντες στη συγκεκριμένη αποστολή. Αυτό το οποίο τίθεται είναι γιατί δεν μπόρεσαν τα μέλη τα οποία πήραν μέρος να συμφωνήσουν στο περιγραφικό κομμάτι της εκθέσεως. Και εγώ δεν πιστεύω στην αναβολή γιατί αυτό θα δημιουργήσει άλλες συνέπειες. Και στο τέλος θα μείνουμε χωρίς έκθεση. Κύριε Κυρία Όκεν, κοιτάξτε, δεν υπάρχουν ε, μόνο κανόνες για την πλειοψηφία και τη μειοψηφία, αλλά οι κανόνες είναι κοινοί για όλους. Τα τρία μέλη της αντιπροσωπείας είναι ισότιμα, παρακαλώ. Αυτό σημαίνει ότι αν υπάρχει μια πλειοψηφία, η πλειοψηφία αυτή θα πρέπει ε, να ληφθεί υπόψη και το ίδιο και η μειοψηφία. Κοιτάξτε, εφόσον παραπέμπετε στους κανόνες, ε, ε, εγώ θα σας δώσω το λόγο όταν το ζητήσετε. Λοιπόν, λέει η Πρόεδρος, ζητήθηκε Ζητήθηκε από τέσσερις βουλευτές, λέει η Πρόεδρος. Uh, με αποχή από πλευρά του κυρίου Μποστινάρου. Όχι, λέει ο κύριος Μποστινάρου. Συμφωνώ με τον Κάσμαν. Uh, the, item can be because of the majority. And uh, in addition... Θα ακυρωθεί το θέμα λοιπόν. Υπάρχει πλειοψηφία για την ακύρωση. Τη διαγραφή εννοεί πρόεδρος. Και σύμφωνα με τους κανόνες όταν μέλη μιας αντιπροσωπείας δεν μπορούν να καταλήξουν σε μια συμφωνία και μιας και η έκθεση για την αποστολή ε, είναι μια απλή περιγραφή του τι είδαν τα μέλη για να μπορέσει η Επιτροπή να εργαστεί σωστά πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Πρέπει να παραδεχτώ ότι το θέμα αυτό δεν αντιμετωπίστηκε με το σωστό τρόπο. Δεν έχει περάσει και πάρα πολύ χρόνος από την αποστολή και με απογοήτευση το διαπιστώνω αυτό. Και σύμφωνα με τις αρμοδιότητες τις οποίες έχω, μπορώ να ζητήσω και να μην υπάρξει έκθεση. Is not able to prepare a report because... Λοιπόν, και να μην υπάρξει έκθεση λοιπόν, διότι τα μέλη μεταξύ τους δεν μπορούν να καταλήξουν. Πέρα από τους αριθμούς στους οποίους έγινε αναφορά, Βέρτμαν, ε, Μπόλαντ και τα λοιπά, εγώ νόμιζα ότι η έκθεση αυτή ήταν το σύνολο των απόψεών σας. Νόμιζα ότι το κείμενο αυτό είχε γίνει ε, με συνένεση μεταξύ σας. Αλλά μιας και δεν συμφωνείτε και εσείς ήσασταν παρούσα, εγώ δεν ήμουν. Και ανάλογα λοιπόν με τις απόψεις τις οποίες ακούσαμε διαπιστώνω ότι δεν καταλήξαμε σε συνένεση, λυπάμαι γι' αυτό και δεν θα συνεχίσουμε τη διαδικασία. Και από εδώ και πέρα ε, το θέμα αυτό παρουσιάζει περισσότερα μειονεκτήματα από όσα πλεονεκτήματα για την Επιτροπή. θα δούμε τι θα κάνουμε με τις αναφορές ε, για που αναφέρονται, που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη ε, αποστολή. Ε, και απλά διαγράφεται το θέμα από την ημερήσια διάταξη. Κατά τα άλλα, πέραν του σημείου αυτού, συμφωνείτε με την ημερήσια διάταξη. Ja, ich möchte nur im Protokoll vermerkt haben, dass äh, unsere Fraktion gegen eine Verschiebung war. Dann bin ich damit einverstanden. Να σημειωθεί όμως ότι η πολιτική μας ομάδα ήταν κατά της αναβολής. Αυτό να σημειωθεί και στα πρακτικά παρακαλώ. Λοιπόν, Επομένως, ελήφθη η απόφαση με... Ελήφθη η απόφαση μόνη αντίθετη γνωμοδότηση της, ε, του ΕΛΚ, της ομάδας του ΕΛΚΑ. Να προχωρήσουμε λοιπόν. Εκτός μικροφώνου, οι, οι διερμήνες δεν ακούν. Α, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, λέει ο κύριος Μποστινάρου. Θα ήθελα να πω ότι κατά την άποψή μου είναι πραγματικά λυπηρό το γεγονός ότι μετά από τόσους μήνες προσπαθειών ε, και δοκιμασιών τελικά δεν καταφέρουμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Ε, ξέρουμε ότι ε, τα μέλη έχουν συνηθίσει σε πολύ δύσκολες και τεταμένες έτσι, αποστολές στις οποίες όμως τελικά καταφέραμε να φτάσουμε σε ένα κοινά αποδεκτό και υπερψηφιζόμενο συμπέρασμα. Αυτό είναι λυπηρό που συμβαίνει τώρα. Ευχαριστώ κύριε Μποστινάρου. Αλλά να προχωρήσουμε. Σημείο 2, έγκριση των πρακτικών τη συνεδριάσεω τη 17η Οκτωβρίου. Έχουμε ε, εγκρίνει την νέα διαδικασία έτσι όπω αυτή έχει συμφωνηθεί από του συναδέλφου συντονιστέ, έτσι ώστε να επιταχυνθούν οι χρόνοι όσον αφορά ε, τα πρακτικά. Τα πρακτικά λοιπόν τώρα μοιράζονται ε, μέσω στις ε, ιστοσελίδες έχουν δημοσιευθεί και επομένως ρωτώ να μάθω εάν υπάρχουν σχόλια ή εάν μπορείτε να αποδεχθείτε τα πρακτικά της 17ης Οκτωβρίου. Κυρία Βέρτμαν για την συνεδρίαση της 17ης Οκτωβρίου. Ευχαριστώ πολύ λέει η κυρία Βέρτμαν. Ε, μετά από την επίσκεψη στην Δανία, μια συναδέλφου των Πρασίνων, είχαμε ε, μια θέση την οποία θα ήθελε να παρουσιάσει. Η θέση αυτή θα έπρεπε θεωρητικώς να φαίνεται στα πρακτικά. Εγώ όμως αντιτίθεμαι σε αυτήν γιατί ε, δεν ήθιστε και αντίθετα από αυτό που είπαν κάποιοι συνάδελφοι, ε, δεν είναι καθόλου συνηθισμένο γραπτή θέση να κατατίθεται απλώς γιατί κάποιος δεν μπορεί να είναι παρόν και να παρίσταται ε, φυσικά εδώ. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ναι, εντάξει, ε, μας ζητήθηκε. Εσείς θέλετε τη δήλωσή σας να την, βάλετε στο, να τη βάλουμε σε παράρτημα. Θέλετε να τη βγάλουμε ή θέλετε να τη βάλουμε σε παράρτημα τη δήλωση που μας εστάλει, λέει η Πρόεδρος. Επιμένω ότι είναι ασύνηθες να δίνεται επεξήγηση ψήφου εφόσον κάποιος σωματικός είναι απόν. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να εισαγάγουμε εδώ έθιμα επειδή κάτι, κάτι βολεύει κάποιον. Είτε είναι κανείς παρόν στην ψηφοφορία και μπορεί μετά να πει κάτι, είτε είναι απόν και τότε δεν μπορεί και δεν θα πρέπει να γίνεται καμιά εξαίρεση. Κοιτάξτε, Εκείνο το πρωί ε, αναγκάστηκα να μπω στο νοσοκομείο και δεν ήμουν ε, παρούσα και απλώς ζήτησα να διαβαστεί η δήλωσή μου. Εντάξει, Νομίζω ότι ούτε ή άλλως είναι πάρα πολύ καλή αναφορά. Δεν ε, πρόκειται να βελτιωθεί με οποιοδήποτε τρόπο, ούτε και με τη δική μου επεξήγηση. Επομένω, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγο να κάνουμε συζήτηση. Πάμε. Πρόεδρος, πολύ ωραία. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ και τη συνάδελφο Ούκεν. Βεβαίως και ε, δεν έγινε με κανένα τρόπο προσπάθεια ε, να παραβιαστούν τα δικαιώματα των υπολείπων συναδέλφων και δι των παρισταμένων στη συνεδρίαση. Εν πάση περιπτώσει θεωρούμε ότι τα πρακτικά έχουν εγκριθεί με αυτήν την τροποποίηση, δηλαδή την διαγραφή της δηλώσεως της κυρίας Όουκεν. Υπάρχουν αντιρρήσεις επί των πρακτικών, όχι άλλες, αντιρρήσεις πολύ ωραία. Όσον αφορά το σημείο 3, ανακοινώσεις της Προέδρου. Θα ήθελα να σας καλέσω να δείτε τις λεγόμενες αμφίβολες ε, αναφορές οι ε, οποίες σας μοιράστηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Ε, μέχρι τώρα δεν έχουμε δει αντιθέσεις ή λοιπές παρατηρήσεις στις συστάσεις που σε αυτές περιέχονται. Επομένως, Ε, αυτό το σημείο θα θεωρηθεί ε, ως ε, σημείο των πρακτικών, θα μπει ως παράρτημα στα πρακτικά και θα θεωρηθεί εγκεκριμένο μαζί με την έγκριση των πρακτικών της σήμερων. Όσον αφορά τώρα την έκθεση, την ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου. Η συγκητής είναι ο κύριος Πάξας, ο οποίος όμως δεν είναι δυνατόν να είναι παρόν ε, και επομένως ε, η Σένστος Εμπράσας ε, θα πάρει το λόγο εξ ονόματός του. Δεν υπάρχουν άλλα θέματα και άλλα σημεία. για την ψηφοφορία για το θέμα της Γαλλικίας να ασχοληθεί παρακαλώ και η ομάδα των συντονιστών. Να δούμε ακριβώς ε, ε, τι έγινε, να ασχοληθούν σήμερα οι συντονιστές με το συγκεκριμένο θέμα. Θα τεθεί στην ε, συνεδρίαση των συντονιστών θα είστε και παρόν και βεβαίως θα συζητηθεί το θέμα και θα ληφθεί η απόφαση από τους συντονιστές. Επί του σημείου αυτό νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο 6, δηλαδή στην κατεξοχήν εργασία μας ε, που είναι να δίνουμε βήμα στους ε, πολίτες. Α, όχι, ζητώ συγγνώμη λέει η Πρόεδρο, ζητώ συγγνώμη. Πέρασα ένα σημείο. Είμαστε στο σημείο 5, γνωμοδότηση σχετικά με την 29η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπα και προηγουμένως, ο συνάδελφος Συμπάρασας θα πάρει το λόγο. Τον θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη, αλλά ο συνάδελφος Πάξας ε, δεν μπορούσε να είναι ανάμεσά μας σήμερα. Έρχεται στις Βρυξέλλες, αλλά αργότερα. Εξ ονόματός του θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνεισέφεραν στην σύνταξη της συγκεκριμένης γνωμοδότησης. Ευχαριστεί λοιπόν ο κύριος Πάξας ε, τους συναδέλφους του. είναι, θα είναι μια πολύ σύντομη παρουσίαση. Τελείωσα. Να ψηφίσουμε τώρα. Θα ακολουθήσουμε λοιπόν τις προτάσεις σας. για την 29η ετήσια έκθεση για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας θέτω σε ψηφοφορία την τροπολογία 1 Βαλένσα. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 2, νέα παράγραφος 1, ε, εμού της ιδείας υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Νέα παράγραφος 1, η τροπολογία 3 Βίλαντ υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Προφορική τροπολογία τώρα. Είναι κάποιος κατά της προφορικής τροπολογίας. Όχι. Λοιπόν, θέτω σε ψηφοφορία ε, την ε, προφορική του Βίλαντ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ζητώ συγγνώμη, πρέπει να επαναλάβω παρακαλώ γιατί βιάστηκα λίγο. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, ποιοι απέχουν. Δεκτή. Τροπολογία 4. Μαντσόνη. Στην παράγραφο 2 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 5. Φερνάντες. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6 Νέα παράγραφος 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 7. Βίλαντ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 8. Ματσόνι. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 10 με 13 ομαδικά, είπε ο κύριος Κάσμαν. Λέει όχι ο κύριος Κάσμαν, λάθος, όχι. Λοιπόν, 9, Βίλαντ. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία, παρακαλώ επανέρχομαι στην τροπολογία 9 Βίλαντ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία στην 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Λοιπόν, προστίθενται οι, οι ψήφοι Βέρτμαν και η δικοί μου. Συνεπώς 5 υπέρ 7 κατά. Απορρίπτεται. Καλά, δεν πειράζει, θα επαναλάβω, λέει η Πρόεδρο, στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Λοιπόν, ψηφίζουμε για την εννέα Βίλαντα. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορία. Εφτά υπέρ 8 υπέρ 8 κατά μία αποχή συνεπώς ε, καταψηφίζεται η τροπολογία. Τροπολογία 10. Γκέριγκερ Ντεόντεμπεργκ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 11. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 12. Όντεμπεργκ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Η 13 τώρα. Ματσόνι. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική παρήθμ 1 στην παράγραφο 5 ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 17 και 18 ταυτόσημες Βίλαν και Μέγερ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές. Η 19 τώρα. Φερνάντες στην 6. Ποιοι είναι υπέρ. Α, όχι, έχει καταπέσει το 19 και το 20 Πηγαίνουμε στην 21 Βίλαντ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Θα υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για την 21. Στην παράγραφο 7. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. 9 υπέρ 6 κατά μία αποχή, συνεπώς γίνεται δεκτή. Γίνεται δεκτή η τροπολογία Βίλαντ. Περνάμε τώρα στην 22, πάντα στην παράγραφο 7 Φερνάντες. Κοιτάξτε, θα ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα και θα δούμε τι θα γίνει με το δεύτερο μετά, λέει η Πρόεδρος. Λοιπόν, το πρώτο τμήμα της 22, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα. Α, όχι, για μια στιγμή. Λοιπόν, το δεύτερο τμήμα έχει καταπέσει πλέον. Περνάμε στην 23, Βαλένσα, ποιοι είναι υπέρ. Α, όχι, και αυτή καταπίπτει, λέει η πρόεδρος εκ των υστέρων. Εφόσον η 21 έγινε δεκτή και η 23 καταπίπτει. Συγγνώμη, αλλά η γραμματεία προ στιγμή δεν μπορεί να με βοηθήσει, λέει η Πρόεδρος. I'm very sorry, some problems with the secretariat. Okay. Έχω ένα μικρό πρόβλημα εδώ. Λοιπόν, 23, 24 και 25 καταπίπτουν ακριβώς γιατί έγινε δεκτή η τροπολογία 21. Περνάμε λοιπόν τώρα στις τροπολογίες 26 και 27, ταυτόσημες Βίλαντ και Φερνάντες. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, ποιοι απέχουν, δεκτές. Τροπολογία 28. Α, όχι, και αυτή έχει καταπέσει. Έχει καταπέσει και 29, φτάνουμε στην 30. 30 Φερνάντες. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία υπαριθμών 30 ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ ψηφίστε Κάρλος ψηφίζεις κι εσύ πέρα της ψηφοφορίας 6 υπέρ 8 κατά Συνεπώς η 30 απορρίπτεται. Τροπολογία 31. Φερνάντες για μια νέα παράγραφο 9. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, ποιοι απέχουν. Δεκτή. Και εδώ ηλεκτρονικός έλεγχος για την 31. Ψηφίζεται. Πέρας της ψηφοφορίας. Λοιπόν, 10 υπέρ 5 κατά, συνεπώς η τροπολογία 31 γίνεται δεκτή. Φτάνω τώρα στην 32 Βίλαντ. Νέα παράγραφο 9, ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, ποιοι απέχουν δεκτή. Προφορική Βίλαντ, είναι κάποιος κατά της προφορικής Βίλαντ, όχι, συνεπώς τίθεται σε ψηφοφορία για μια νέα εννέα. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, ποιοι απέχουν δεκτή. Τροπολογία 33. Φερνάντες ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 33. Πέρα της ψηφοφορίες. 9 υπέρ. 6 κατά μία αποχή. Η 33 γίνεται δεκτή. Φτάνουμε στην 34 στην παράγραφο 10. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν δεκτή. Τροπολογία 35 Βίλαντα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 36 Φερνάντες. Ποιοι είναι υπέρ. <clears throat> κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 37 Βίλαντα. Νέα παράγραφος 13. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 38 στην 14. Φερνάντες. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 39 Βαλένσα 14. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία υπαριθμών 40 Βίλαντα στην παράγραφο 15 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 Φερνάντες στη 15 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή 42 Γκέριγκελ Ντέοντεμπεργκ νέα παράγραφος 15 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 44 Φερνάντες στην 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 43 Μπέκερ ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 45 Μέιερ στην 17 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 46 Ödenberg. Νέα παράγραφος 17. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Θέτω σε ψηφοφορία την 46. Πέρα της ψηφοφορίας. 4 υπέρ. 8 κατά τέσσερις αποχές. Απορρίπτεται. Θέτω σε ψηφοφορία τώρα το σύνολο του ψηφίσματος. Ποιοι είναι υπέρ. Πέρα της ψηφοφορίας 14 υπέρ, 1 κατά, 0 αποχές, η έκθεση γίνεται δεκτή. Ευχαριστούμε λοιπόν τον συνάδελφο Πάξας όπως και τον συνάδελφο Ιμπράξας. Περνάμε στο σημείο 6 λοιπόν. Περνάμε στις τροπολογίες 749 ε, ε, ε, Βρετανών υπηκών που δεν είναι παρόντες και γι' αυτό δίνουμε απευθείας το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, eh, για τις αναφορές του σημείου 6, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Um, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρόκειται για την χρήση σε βρετανικά αεροδρόμια σαρωτών σώματος. Τον Νοέμβριο του 2011 η Κομισιόν ενέκρινε κανονισμό που επιτρέπει τη χρήση σαρωτών ασφαλείας σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια που χρησιμοποιούν κύματα χιλιοστού ενώ δεν επιτρέπονται αυτοί που χρησιμοποιούν ακτίνες χ. Προβλέπεται επίσης από τον κανονισμό και το λεγόμενο opt-out, δηλαδή ο επιβάτης μπορεί να ζητήσει εναλλακτική μέθοδο ε, έρευνας. Το Δεκέμβρη του 2011 το Ενωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε, κοινοποίησε μάλλον στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν εγκρίνει το opt-out και όποιο αρνείται να περάσει από το security scanner δεν μπαίνει στο αεροπλάνο. Ως follow-up προβήκαμε σε νομική αξιολόγηση με βασικό ερώτημα εάν εκείνο το no scan, no fly του Ηνωμένου Βασιλείου αποτελεί παραβίαση του ευρωπαϊκού κανονισμού όπως ισχυρίζονται οι αναφέροντες ή εάν υπάρχει περιθώριο και το ανέχεται ο κανονισμός. Η νομική μας αξιολόγηση κατέδειξε και πιστεύουμε ότι το Βρετανικό μέτρο αποτελεί παραβίαση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Ξεκίνησε λοιπόν η, διαδικασία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία διαδικασία προ-προσφυγής για παραβίαση και τον 22 Νοεμβρίου το Ενωμένο Βασίλειο εξέδωσε νέα οδηγία προς τα αεροδρόμια που αντικαθιστά την no scan no fly αυτή πολιτική. Επομένως οι επιβάτες τώρα επιτρέπεται να ζητήσουν και να λάβουν εναλλακτική μορφή έρευνα. Άρα τελικά το Ενωμένο Βασίλειο δέχθηκε την ε, νομική αξιολόγηση της Επιτροπής, αντικατέστησε την no-fly πώληση. Υπάρχει τώρα και δεύτερο επιχείρημα για το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ, διότι υπάρχουν παλαιές μηχανές ε, που χρησιμοποιούν ε, ακτίνες χ και είναι επομένως ε, μικρότερες από 20 κύματος χιλιοστού. Αυτές όμως αντικαταστάθηκαν ήδη εδώ και ένα χρόνο. Λοιπόν, η αναφορά που έγινε από τους πολίτες που στράφηκαν στην Επιτροπή μας όχι απλά ήταν ε, τεκμηριωμένη και έγινε ακριβώς αποδεκτή και από τις εθνικές αρχές. και πρέπει να υπάρξει σεβασμός των ευρωπαϊκών ρυθμίσεων. Πέραν αυτού τώρα, ο συνάδελφος Μποστινάρου έχει ζητήσει το λόγο. Ε, Επιτρέψτε μου κυρία Πρόεδρε, και νομίζω ότι μιλώ και εξ ονόματος όλων των συναδέλφων, δείχνει αυτό τόσες φορές πόσο αποτελεσματική είναι η Επιτροπή Αναφορών και πόσο σημαντικό και ευεργετικό ρόλο παίζουμε υπέρ του Ευρωπαίου πολίτη. Κατορθώνουμε έτσι να βραχύνουμε τις διαδικασίες, εντοπίζοντας τα προβλήματα εκεί όπου βρίσκονται και βεβαίως με τη συνεργασία και ε, στράτευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία επιθυμώ να ευχαριστήσω. Ευχαριστώ κύριε Μποστινάρου. Θα ενημερώσουμε τον υπογράφοντα και θα τον ευχαριστήσουμε γιατί μας έδωσε τη δυνατότητα να εντοπίσουμε μια, μια μη σωστή ε, αντιμετώπιση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και φέραμε εις πέρα στην αποστολή μας νομίζω με μεγάλη ταχύτητα και επιτυχία. Μπορούμε να κλείσουμε λοιπόν την αναφορά θετικά. Περνάμε στην επόμενη αναφορά, την αναφορά που παρουσιάζει, που καταθέτει Βρετανός πολίτης εξ ονόματος των λεκτόρων ξένης γλώσσας στα ανώτατα ιδρύματα της Ιταλίας και τις διακρίσεις που υφίστανται. Ο υπογράφων έχει το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη. Το προηγούμενο έτος συζητήσαμε ε, το άρθρο 26 του νόμου Τζεμέλη και υπήρχε κάτι στη διατύπωση του συγκεκριμένου νόμου που έπρεπε να, ε, να εξετάσουμε προσεκτικά και να δούμε και πώς ε, είχε εφαρμοστεί στην πρακτική. Άφησα στη γραμματεία τρεις γνωμοδοτήσεις για τον συγκεκριμένο νόμο που διευκρίνιζαν ότι δεν έπρεπε να διακόψει τη διαδικασία ο νόμο, ε, εναντίον του νόμου Τζελμίνη. Ο νόμος Τζελμίνη ε, είναι εν μέρη συμβατός με την κοινοτική νομοθεσία Υπήρξαν 17 περαιτέρω σελίδες ε, αποδεικτικών στοιχείων και ζητήσαμε μία συνάντηση ε, ε, έτσι ώστε να βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κοιτάξτε τις σημερινές εφημερίδες για να δείτε ότι η Ευρώπη πράγματι είναι στην κρίση και η μετανάστευση και η ελεύθερη διακίνηση είναι ένα θέμα πάρα πολύ καυτό. Οι εθνικές κυβερνήσεις γνωρίζουν ότι αν απομακρυνθούν από την κοινή γνώμη θα χάσουν την εξουσία. Ο Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου Λίντινγκτον που ζήτησε να με συναντήσει την Πέμπτη επανειλημμένα, θαραλέα και με ειλικρίνεια κατήγγειλε τη συμπεριφορά της Ιταλίας ως ανήθικη και παράνομη και τώρα μπορεί να μεταφέρει κάποια ενθαρρυντικά στοιχεία από τους Ιταλούς Υπουργούς Καρότσα και Μπονίνο. Ε, η Βρετανική Πρεσβεία, η Ισπανική, η Ιρλανδική, η Γερμανική και η Γαλλική έχουν αρχίσει και ενδιαφέρονται και συνεργάζονται ε, στην Ρώμη. Ε, όχι με έμεσο τρόπο, αλλά άμεσα και καθαρά η κυβέρνηση του Σίλβιο Σκόνη πέρασε το νόμο Τζελμίνη με δεδομένο των στόχο... και αυτό φαίνεται στα πρακτικά της Ιταλικής Γερουσίας υπαριθμών 94 του Δεκεμβρίου 10 λέγοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ε, ε, λαμβάνονται αποφάσεις εις βάρος των συμφερόντων των ιδίων των πανεπιστημίων. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο νόμος αυτός είναι η κορονίδα θα έλεγα ή ο πρόδρομος μάλλον της ε, επερχόμενης κοινότητας ε, χωρίς νόμο, με διακρίσεις, με ρατσισμό. Στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι τα πράγματα, πρόκειται για μια δικτατορική επιβολή θέσης. Αν πετύχει αυτή η διαδικασία, αυτό σημαίνει ότι μετά από 30 χρόνια συζητήσεων δεν μπορεί να εφαρμοστεί ισότιμα η ενιαία αγορά. Οι κανονικοί τίμοι κατά τα άλλα μετανάστες καθηγητές, ε, κανένας δεν μας κατηγόρησε ότι είμαστε απατεώνες οι τουρίστες του τομέα της υγείας ή της ευημερίας και παρότι πετύχαμε έξι αποφάσεις από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ακριβώς επειδή τις πετύχαμε υφιστάμεθα την άδικη επιβολή άποψης. Κοιτάξτε στον ε, φάκελο, θα δείτε εκθέσεις των εμπειρογνωμόνων από καθηγητές ε, και από ανώτατους δικαστικούς. Θα δείτε να χαρακτηρίζεται η ρύθμιση Τζελμίνη απαράδεκτη, υπονομευτική της εξουσίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, της αρμοδιότητας συγγνώμη, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ο καθηγητής Νόριν Μπάροους λέει το να κλείσει ο φάκελος αυτός είναι ένα μήνυμα στην Ιταλία και όλα τα κράτη-μέλη ότι η συστηματική περιφρόνηση των θεμελιωδών ευρωπαϊκών κανόνων είναι κάτι το οποίο τελικά θα επικρατήσει. Εν τω μεταξύ δικαστήρια στο Λέτσε, το Τωρίνο, το Μιλάνο, την Πρέσια αναδρομικά έχουν αρχίσει και σβήνουν κάποιες περιπτώσεις ε, δικαστικών αποφάσεων. 60% μειώθηκαν οι μισθοί στην Κατάνια, το Σαλέντο και το Μπέργαμο επί τη βάση του νόμου Τζελμίνη που επηρεάζει άμεσα μόνο τους μη Ιταλούς λέκτορες. Πραγματικά ένας καθαρά ρατσιστικός νόμος. Λοιπόν, θα πρέπει να επικρατήσει η άποψη του Υπουργού Λίντιγκστον, αλλά αλλιώ φοβάμαι ότι θα μας καταπιεί όλους η καταχρηστική αντίληψη για την Ευρώπη του κυρίου Μπερλουσκόνη και των ομοίων του. Ευχαριστώ πολύ και εσάς. And now, where's the other one? Uh, does Mr. Innes want to say something? Mr. Innes. There is even Mr. Innes. Είναι και ο κύριος Ίνες εδώ. Θέλετε να προσθέσετε κάτι, όχι. Φρανθίσκο Πέρες Φλόρες από την Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που, έδωσε, που έστειλε στην Επιτροπή σας, ε, η Επιτροπή αναφέρεται στην ανάλυση η οποία ε, έλαβε χώρα μετά από τις σχετικές πληροφορίες που μας έστειλαν οι Ιταλικές Αρχές για τον νόμο Τζελμίνη. Ο, ο, αναφέρον, ο αναφέρον επίσης έστειλε επιπλέον ε, πληροφορίες ε, τις οποίες συγκρίναμε με αυτά τα στοιχεία τα οποία είχαμε τελευταία φορά τον Ιούλιο του 2013. Έκαναν αξιολόγηση οι υπηρεσίε της Κομισιόν ε, των πληροφοριών που έλαβαν και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι δεν έχουμε στοιχεία ε, τα οποία θα οδηγήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει διαδικασία επιπαραβάση κατά της Ιταλίας. Επίσης, το Σεπτέμβριο τρέχοντος έτους εμείς κοινοποιήσαμε εις τον αναφέροντα την πρόθεσή μας να κλείσουμε την διαδικασία πριν κλείσουμε το φάκελο, δώσαμε την δυνατότητα στον αναφέροντα να δώσει ενδεχόμενες επιπλέον, ισχυρές, ε, ε, επιπλέον ισχυρά στοιχεία, έτσι ώστε να τροποποιήσουμε την αρχική μας θέση. Όπως είπε ε, και ο αναφέρον, έστειλε περαιτέρω παρατηρήσεις μαζί και με άλλα σχόλια και αποδεικτικά στοιχεία την 14η Νοεμβρίου. Αυτά τα στοιχεία τα αναλύουμε τώρα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 το βάρος της απόδειξης για οποιαδήποτε περίπτωση διαδικασίας επιπαραβάσης εναντίον οποιαδήποτε κράτους ε, μέλους είναι στα χέρια της Επιτροπής. Θα θυμάστε επίσης ότι η Κομισιόν ξεκίνησε διαδικασία επιπαραβάση κατά της Ιταλίας που οδήγησε στην ετοιμιγορία του ε, δικαστηρίου του Ιουλίου 2006 ε, όπου το δικαστήριο απεφάνθη ότι η Ιταλία έπρεπε να ε, δώσει στοιχεία έτσι ώστε να ε, σταματήσει τη διαδικασία επί παραβάση η Κομισιόν. Ε, όμως τώρα φτάσαμε στο συμπέρασμά μας. Πρόθεσή μας είναι να κλείσουμε τον φάκελο βάσει αυτών των στοιχείων που θα σας αναφέρω τώρα. Πρώτα απ' όλα, ο αναφέρον αναφέρει ότι οι λέκτορες, τότε λετόροι στα Ιταλικά, δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες, καθώς επίσης και τα ίδια δικαιώματα, τα οποία έχουν αντίστοιχα οι Ιταλοί εργαζόμενοι που καλύπτουν παρόμοια θέσεις. Επίσης, ε, διατείνεται ότι θα έπρεπε να ε, ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία τους με αύξηση 2,5% για κάθε χρόνο, ε, καθώς επίσης και μία αύξηση 6 μισθών επί τη βάση υπολογισμού 8% για κάθε χρόνο υπηρεσίας. Μας έχει δώσει ο αναφέρον πίνακες που δείχνουν τι ακριβώς μισθό κερδίζουν αυτή τη στιγμή οι λέκτορες. Εμείς Είπαμε στον ε, ε, αναφέροντα ότι δεν έχουμε στοιχεία ότι οι πίνακες αυτοί διαφέρουν από τους πίνακες που ισχύουν για άλλους Ιταλούς εργαζόμενους ε, σε ίδιες θέσεις ή παρόμοιες θέσεις. Επομένως, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε διαδικασία επιπαραβάση βάσει του άρθρου 45 της συνθήκης. Επιπλέον, ο αναφέρον ε, ε, διατείνεται ότι η συνέχιση της, ε, της καριέρας των πρώην ελετόρι και εφεξής CES δεν έχει προχωρήσει κανονικά. Επίσης διατείνεται ότι αντιτίθεται στις ετοιμιγορίες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου η πράξη η οποία ισχύει στην η πρακτική συγγνώμη, η οποία ισχύει στην Ιταλία. Ε, αυτός ο διαχωρισμός ε, δηλαδή αντιτίθεται στις μέχρι τούδε αποφάσεις ε, του δικαστηρίου. Επίσης διατείνεται ότι για τους Ιταλούς εργαζόμενους δεν ισχύει αυτού του είδους ο διαχωρισμός βάσει του νόμου του 1995 δεν θεωρούμε ότι ε, δεν, ε, ε, ότι δεν πρέπει να υπόκεινται στις συλλογικές διαδικασίες οι μη Ιταλοί, Ευρωπαίοι εργαζόμενοι. Επίσης, δεν φαίνεται σαφώς ότι ο νόμος Τζελμίνη είναι υπεύθυνο για αυτήν την πάυση ή την παρεμπόδιση της καριέρας, αλλά μάλλον ο αρχικός νόμος του 95. Τρίτον, ο αναφέρον διατείνεται ότι η τελευταία φράση του 26 παράγραφος 3 του νόμου Τζελμίνη αναφέρεται σε παραβίαση πολλών συμφωνημένων και επικυρωμένων διεθνών συνθήκων όπως ας πούμε το άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Επιπλέον, οι αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων ε, ε, είναι αποφάσεις οι οποίες μπορούν να εφεσιβληθούν. Επομένως, από τη στιγμή που δεν υπάρχει διαφορετική ερμηνεία του νόμου, δεν μπορεί η Κομισιόν να ε, τεκμέρει ότι υπάρχει εδώ παραβίαση του άρθρου 45 της, των Συνθήκων Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως δεν μπορεί να αλλάξει η απόφαση της Κομισιόν βάσει των στοιχείων της 14ης Νοεμβρίου. Θα συνεχίσει πάντως η Κομισιόν την εν λόγω ανάλυση. Ευχαριστώ. Η κυρία Όκεν. Sorry. Øh, det er blot fordi, altså jeg sidder her, jeg har kendt til de her sager. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι πρόκειται για μια υπόθεση που παρακολουθούμε επί πολλά έτη. Έχουμε και άλλους που έχουν εργαστεί στην Ιταλία και πληρώνονταν λιγότερο. Εγώ έχω προετοιμαστεί, διάβασα και την απάντηση της Κομισιόν, η οποία λέει ότι θα λάβουμε και άλλες προφορίες αργότερα. Αλλά αυτό δεν αρκεί πριν να κλείσουμε την αναφορά πρέπει να δούμε όλες τις απαντήσεις. Εδώ μαθαίνουμε νέες πληροφορίες. Είναι δύσκολο να μπορέσω να αποφασίσω στην βάση αυτής της πολύ σύντομης τοποθέτησης της Κομισιόν για το αν είναι δικαιολογημένη ή όχι η ε, αναφορά. Πρέπει τουλάχιστον να έχουμε το χρόνο να ξαναδιαβάσουμε το φάκελο, να δούμε τι ακριβώς έχει λεχθεί από κάθε πλευρά δεν ακούω τουλάχιστον από αυτά που άκουσα δηλαδή, δεν, δεν διακρίνω να έχει βρεθεί κάποια λύση. Και αυτά που λέει τώρα η Κομισιόν, γιατί δεν μας τα έχει διαβιβάσει εκ των προτέρων. Διαβάζω εδώ ότι η Κομισιόν θα μας ενημερώνει. Μα τι μας ενημέρωσε, παρόλο που το λέει. Το έχουν γράψει, αλλά δεν το έκαναν. Δεν το έπραξαν. Και γι' αυτό θεωρώ ότι πρόκειται για απώλεια χρόνου. Ο κύριος Μποστινάρου. Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Δύο παρατηρήσεις έχω. Είναι προφανές ότι η απάντηση της ε, Επιτροπής, της Κομισιόν δεν επαρκεί. Πρώτα διακρίνω μια αντίφαση στους όρους. Από τη μια μεριά λένε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις κάποια διακριτική μεταχείρισης σε βάρο του αναφέροντος, ταυτόχρονα όμως επιβεβαιώνουν ότι δεν έχουν και επίσημο κατάλογο των αμοιβών για τους Ιταλούς, των μισθών για τους Ιταλούς και, για το, και των μισθών για τους λέκτορες. Αν αυτό συμβαίνει, είναι δύσκολο διότι στο κάτω της γραφής είμαστε στο 2013. Κάθε στοιχείο που έχει σχέση με τα μισθολόγια των πανεπιστημίων είναι δημόσιο στοιχείο. Μπορεί εύκολα να βρεθεί σε κάθε χώρα μέλος. Μάλιστα και ακόμα και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί είναι τόσο δύσκολο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντοπίσει το μισθολόγιο των πανεπιστημίων και να δει αν από εκεί προκύπτουν κάποιες ενδείξεις ή όχι. Μα είναι πραγματικά κρυσταλλίνη το επιχείρημα. Τότε μόνο θα μπορέσει να κρίνει εάν είναι, αν στερείται θεμελίων η αναφορά. Έχοντας λοιπόν υπόψη αυτό το γεγονός, θα προτείνω η αναφορά να παραμείνει ανοιχτή και από την πλευρά της Κομισιόν να λάβουμε μια ξεκάθαρη απάντηση με αποδεικτικά στοιχεία, διότι εν τέλει, βέβαια, το πλέον ε, από χρόνο αποδεικτικό στοιχείο είναι το μισθολόγιο. Αυτό δείχνει εάν υπάρχει ίση, ισότιμη μεταχείριση και ισότιμη αμοιβή για ίση εργασία. Και αν δεν Στη βάση αυτή θα αποφασίσουμε τότε αν θα κλείσουμε την αναφορά. Αλλά όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, εγώ προτείνω να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και να ζητήσουμε από την Κομισιόν να προβεί σε μια κρίση βασισμένη σε στοιχεία και όχι σε ερμηνείες. Πρόεδρος, θέλουν άλλοι συνάδελφοι να πάρουν το λόγο. Όχι, θα δώσω επομένω ξανά... Ε, α, υπάρχει ένας συνάδελφος που θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, συνειδητοποιούμε εδώ ότι το θέμα των αμοιβών είναι πολύ ευαίσθητο θέμα. Εάν η Κομισιόν δεν μπορεί να είναι σαφής ε, και δεν έχει τα στοιχεία που θα τις επιτρέψουν να ε, είναι σαφείς, θα πρέπει να έχει το χρόνο να αξιολογήσει περαιτέρω τα στοιχεία της αναφοράς αυτής, έτσι ώστε να μας δώσει απάντηση τεκμηριωμένη επί στοιχείων. Ε, ευχαριστώ πολύ. Θα δώσουμε το λόγο τώρα στον αναφέροντα ένα λεπτό για την απάντησή σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Μπορώ μόνο να επαναλάβω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία. 60% περικοπές μισθών είχαμε ε, και όλα τα αποδεικτικά στοιχεία περί αυτού τα ε, έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, και επίσης έχουμε όλα τα στοιχεία τα οποία μας έχει απαντήσει ο Επίτροπος ή το γραφείο του Επιτροπή Επιτρόπου Άντερς και νομίζω ότι υπάρχουν και όλα τα στοιχεία μάλιστα στα αγγλικά. Ε, θα ήθελα να υποβληθούν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία έχω υποβάλει ε, σε έκθεση πραγματογνωμοσύνης έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε κάποιο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ λέει η Πρόεδρος. Νομίζω ότι τώρα είναι σαφέ, ότι θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά εν αναμονή περαιτέρω σχολείων από πλευρά τη Ευρωπαϊκή επιτροπή, ε, η οποία θα έχει μελετήσει εντωμεταξύ τα πολυπληθή έγγραφα τα οποία έχει στείλει ο αναφέρον στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να διευθετηθεί το ζήτημα των λεκτόρων, καθηγητών ξένων γλωσσών στην Ιταλία, ένα πρόβλημα ανοιχτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το οποίο, το οποίο συγγνώμη, ακόμα δεν έχει βρει λύση θα ήθελα και εγώ να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν είναι δυνατόν ε, ταχύτατα να μας ε, δώσει απάντηση έτσι ώστε και εμείς με τη σειρά μας ε, να απαντήσουμε στον αναφέροντα. Θέλει κάποιος άλλος αναφέρον να πάρει το λόγο. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Όχι. Συμφωνείτε με τον προναλήσαντα και τον στηρίζετε. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε. Επομένως, παραμένει ανοιχτή αυτή η αναφορά ε, και ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ε, ε, κοινοποιήσει την απόφασή της μετά από έλεγχο των στοιχείων. Ευχαριστούμε τους αναφέροντες που ήταν και παρόντες και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως. Πρόκειται για το σημείο 8, αναφορά 1954 του 2012 που έχει υποβληθεί από τον ε, η, ε, Ουγγρικής Ιθαγένειας πολίτη Φαζάκα Πάλμα με δύο υπογραφές σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση της οδηγίας από πλευρά σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών τίτλων των ΜΕΟΝ. Έχουμε εδώ ε, παρουσία των αναφέροντων και έχουμε επομένως τον κύριο Φαζάκας. La parola a Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω όμως ότι κανονικά δεν πρέπει να λάβω εγώ το λόγο πρώτος. Έτσι δεν είναι. Πρώτα είναι το σημείο 8. I was another mistake. Okay. Mrs. Bodrogi. Η κυρία Μποντρότζη. Okay. So my name is Bea Bodrogi. I'm a human rights lawyer from Hungary. Είμαι δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Ουγγαρία και εκπροσωπώ και μάλιστα τρεις μη κυβερνητικές οργανώσεις. στην αναφορά μας θεωρούμε ότι η Ουγγαρία δεν έχει συμμορφωθεί ε, με τις ε, διατάξεις οδηγίας 2005-36 της Ευρωπαϊκής ε, Κοινότητας σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών τίτλων των ΜΕΟΝ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να αναφερθώ ε, στην σημασία αυτής της αναφοράς. Από τη μία μεριά έχουμε την οδηγία η οποία αναφέρεται στην αναγνώριση επαγγελματικών τίτλων των μεών ε, και γενικότερα στην ε, επαγγελματική αυτονομία και ανεξαρτησία των ιδίων. Από την άλλη πλευρά σχετίζεται με τις γυναίκες οι οποίες θέλουν να ξέρουν πώς, πότε και με ποιον τρόπο και παρουσία τίνος θέλουν ε, να γεννήσουν. Ε, τα συστήματα, ε, τα ιατρικά στην Ουγγαρία βασίζονται κυρίως στην παρουσία του γιατρού. Ωστόσο, η διαδικασία της, του τοκετού, η διαδικασία της γέννησης είναι κάτι διαφορετικό και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη πολλά διαφορετικά στοιχεία που δεν μπορεί όλα να τα καλύψει ο γιατρός. Εμείς ουδόλως αμφισβητούμε το ρόλο των γιατρών. Ωστόσο, η επιβίωση πολλών ε, γυναικών και πολλών νεογέννητων παιδιών ε, ε, οφείλεται στην προώθηση της ιατρικής τεχνολογίας. Είναι γεγονός ότι η παρουσία του γιατρού μπορεί να βοηθήσει στις περισσότερες περιπτώσεις. Ωστόσο, η παρουσία των μεών είναι πάρα πολύ σημαντική. Έξι στις δέκα γυναίκες έχουν υποστεί σαρική τομή κατά τη διάρκεια του, του τοκετού. Επίσης είναι πολλές οι γυναίκες οι οποίες λαμβάνουν την στιγμή του τοκετού τους ιατρικές παροχές τις οποίες δεν θα ήθελαν ε, θεωρούμε λοιπόν ότι ε, και για να αυξηθεί και ο αριθμός των γεννήσεων θα πρέπει να αλλάξει το σύστημα. Στην Ουγγαρία είναι πάρα πολύ ε, ακριβώς ο τοκετός και θεωρητικός όμως καλύπτονται τα έξοδα από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι ε, γυναίκες παρακολουθούνται ε, σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους ε, και προσπαθούν να τις παρακολουθεί ο ίδιος γιατρός έτσι ώστε να φτάσουν στη στιγμή του τοκετού έχοντας περισσότερες ελπίδες να έχουν την σωστή αντιμετώπιση. Η σημασία των μεών έχει υπογραμμιστεί σε πολλές εκθέσεις. Τα Ηνωμένα Έθνη στην ε, αναφορά τους ε, ε, για, τα έτη 11 και 12 αναφέρουν ότι η παρουσία των μεών είναι ιδιαίτερα σημαντική τη στιγμή των τοκετών. Επίσης, ε, η παρουσία των επαγγελματιών μεών μειώνει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ε, τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει η υγεία και η ζωή των νεογέννητων και των ε, μητέρων τους στο, ε, στην παράγραφο 42 της οδηγίας 2005 αναφέρονται, ε, αναφέρεται ότι οι ΜΕΕΣ μπορούν πέρα από την παρουσία τη στιγμή του τοκετού ε, να βοηθήσουν τις εγκυμονούσες στη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους στους τακτικούς και περιοδικούς ελέγχους. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεργασία ανάμεσα στις ΜΕΕΣ και τους ε, γιατρούς. Ε, και βεβαίως είναι εξίσου σημαντικό οι γυναίκες να έχουν την δυνατότητα να αποφασίζουν για το κατά πόσον, για το κατά πόσον ε, ζητούν την παρουσία ΜΕΑΣ στη διάρκεια του τοκετού Πολύ ε, περισσότερες γυναίκες ε, πλέον επιθυμούν τις, ε, την παρουσία των μεών τη στιγμή του τοκετού, ακόμα και χωρίς την παρουσία γιατρού, ενώ σημειώνεται βεβαίως ότι αυτό είναι δυνατό μονάχα σε φυσιολογικές εγκυμοσύνες και επομένως εγκυμοσύνες χωρίς πρόβλημα η εσφαλμένη εφαρμογή ή η μη συμμόρφωση του άρθρου 42 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2005 από την Ουγγαρία δεν δίνει την προβλεπόμενη ανεξαρτησία στις ε, ε, ΜΕΕΣ ούτε δίνει στις ΜΕΕΣ την δυνατότητα να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους, τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες εντός και εκτός των νοσοκομείων. Στην Ουγγαρία 99% των γυναικών ε, προτιμούν, ε, επιλέγουν το νοσοκομείο για τον ε, τοκετό και το σύστημα στην Ουγγαρία σχεδόν αποκλειστικά προβλέπει τον γιατρό, τον γυναικολόγο για τη στιγμή του τοκετού. Ε, θεωρούμε ότι αυτό δεν, δεν προβλέπεται ακριβώς από την οδηγία. Ε, όσον αφορά τώρα την... Ε, την ευθύνη και ιατρικά, δηλαδή επιστημονικά και απέναντι στο δίκαιο είναι ο γιατρός. Αυτό όμως οδηγεί καμιά φορά σε αδικαιολόγητες παρεμβάσεις. Τώρα η κυβέρνηση επιτρέπει στις ΜΕΕΣ να πηγαίνουν και σε γεννήσεις εκτός ιδρυμάτων. Υπάρχει όμως το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει αποφασίσει κατά της Ουγγαρίας σε μια υπόθεση. Ενημερώνουμε επίσης την Επιτροπή σας ότι η Ουγγρική κυβέρνηση ξεκίνησε συζήτηση για την τροποποίηση των ισιών των κανονισμών για την φροντίδα της μητρότητας έχουν αποσταλεί σχέδια για τις τροποποιήσεις αυτές σε επαγγελματικέ οργανώσεις και οι τρεις οργανώσεις ωστόσο που έχουν υπογράψει τη σημερινή αναφορά έχουν υποβάλει το σχετικό υλικό στο αρμόδιο Υπουργείο. Έχουμε αναγνωρίσει λοιπόν τις προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση όσον αφορά την επέκταση των αρμοδιοτήτων των μεών για να συμμετέχουν μόνες τους ανεξάρτητα δηλαδή σε γένες χωρίς ετοκετούς που δεν ε, ενέχουν κίνδυνο αλλά μέχρι τώρα τα σχέδια της κυβέρνησης δεν ε, συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Εξακολουθούν να επιμένουν ότι μόνο ο γιατρός έχει το δικαίωμα να κρίνει ποιος το είναι χαμηλού κινδύνου ή υψηλού κινδύνου και να αποφασίζει αν η έγκυος ε, θα εισαχθεί στο νοσοκομείο. Εν τέλει, αυτά μειώνουν την ανεξαρτησία και αυτονομία των μεών. Εμείς πιστεύουμε ότι οι ΜΕΕΣ και οι γιατροί πρέπει να συνεργάζονται με αμοιβαία εμπιστοσύνη και ε, σεβασμό. Αλλά αυτά δεν μπορούν να εξασφαλιστούν με την αναθεώρηση που προτείνει η κυβέρνηση και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάθει μεγάλες ζημίες από την ιστορία αυτή. Εμείς οι γυναίκες πρέπει να ξεκινήσουμε τις αλλαγές. Ελπίζω ότι η αναφορά μας θα αποδειχθεί σημαντική και ότι αποτελεί ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση της αλλαγής. Παρακαλούμε την Επιτροπή σας να μην κλείσει το θέμα, να μην απορρίψει την αναφορά μας και να λάβει τα μέτρα που θα κρίνει απαραίτητα για να συμβάλλει ώστε να επιτευχθούν οι αλλαγές που επιζητούμε. Ευχαριστώ. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Λαμβάνει το λόγο ο κύριος Ζίγμουντ. Thank you, uh, uh, Actually, my... Ευχαριστώ. Λέγομαι Κωνσταντίνος Τομαράς. Είναι σημαντικό το θέμα. Γιατί φέρνει σε επαφή δύο σημαντικά συστήματα αφενός τα εθνικά συστήματα υγείας και τον τρόπο οργάνωσής τους και λειτουργίας τους και το, το φέρνει σε επαφή με τους κανόνες της Ένωσης για τα επαγγελματικά προσόντα. Όπως είπε ήδη αναφερομένη, οι κανόνες αυτοί προβλέπουν ειδικέ ρυθμίσεις για τις ΜΕΕΣ. Λίγα βασικά τώρα σχόλια, για, περισσότερο για διευκρίνηση. Η ΜΕΑ είναι ένα επάγγελμα το οποίο ευεργετείται από την αυτόματη αναγνώριση, καθεστώς αυτόματης αναγνώρισης που αποκαλούμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή υπάρχει εναρμόνιση των ελαχίστων απαιτήσεων σε όλες τις χώρες μέλη. Και αυτό στη βάση της οδηγίας επαγγελματικών προσόντων. Αυτό σημαίνει ότι στην πράξη οι ΜΕΕΣ σε ολόκληρη την Ευρώπη οφείλουν να πληρούν τα ίδια ελάχιστα στάνταρτ ετών εκπαίδευσης, εμπειρίας κλπ. Ωστόσο είναι μια ειδική κατηγορία αυτόματης αναγνώρισης μές με την έννοια ότι η οδηγία προβλέπει κάποιες δραστηριότητες που θα πρέπει να μπορεί να ασκεί σε κάθε χώρα μέλος το επάγγελμα. Μεταξύ αυτών των δραστηριοτήτων είναι ορθό να λεχθεί όπως είπε και αναφερομένη η διάγνωση τοκετών και παρακολούθηση και συνοδεία ε, ομαλών τοκετών. Αυτές είναι οι δραστηριότητες που θα πρέπει να μπορούν να ασκήσουν οι ΜΕΕΣ. Ίσως να σας ενδιαφέρει ακόμη να ακούσετε ότι έχουμε τροποποιήσει πρόσφατα την οδηγία και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τα οποία όργανα συμφώνησαν. Η νέα έκδοση της οδηγίας αυτής θα δημοσιευτεί ε, τον επόμενο χρόνο. Κάποια θέματα άλλαξαν για τις ΜΕΕΣ αλλά όχι αυτό περί δραστηριοτήτων. Η νομοθεσία λοιπόν όσο έχει τώρα έτσι θα συνεχίσει να έχει και στο μέλλον. Ενώ λοιπόν τώρα είναι ορθό να πει κανεί ότι η οδηγία προβλέπει προσόντα και δραστηριότητε, οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι κάθε χώρα μέλος οργανώνει το δικό της σύστημα υγείας με το δικό της τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές παραδόσεις κλπ. Εκεί λοιπόν είναι το σημείο τομή των δύο συστημάτων και εκεί φαίνεται να ε, προκαλείται το πρόβλημα. Αυτό που προτιθέμεθα εμείς να κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, το έχουμε θέσει υπόψη του Κοινοβουλίου, άλλωστε είμαστε σε επαφή με τις Ουγγρικές Αρχές για να δούμε πού ακριβώς έχουν σχεδιάσει το σύστημα και ιδίω εν ώψη και του νέου νόμου που συντάσσεται για να δούμε μήπως υπάρχει κάποια παρανόηση σχετικά με το περιεχόμενο του νόμου και πώς αυτός ε, δρά σε σχέση με την οδηγία μας. Η Ουγγαρία θεωρεί η αναφερομένη ότι δεν έχει εφαρμόσει ορθά την οδηγία περί επαγγελματικών προσόντων. Και γι' αυτό είναι το σημαντικό να πούμε ότι μιλούμε εδώ για την αλληλεπίδραση δύο συστημάτων διότι εμείς ελέγξαμε τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζει την ίδια την οδηγία η Ουγγρική κυβέρνηση και εδώ δεν βλέπουμε κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα φαίνεται να εντοπίζεται ε, στον τρόπο με τον οποίο οργανώνουν τις αρμοδιότητες και ευθύνες εντός του δικού τους συστήματος υγείας. Γι' αυτό όμως θα χρειαστεί να δούμε πώς το έχουν κάνει και όπως είπα να δούμε και τι θα προβλέπουν οι νέες ε, διατάξεις τους το μόνο που μπορώ να πω για την ώρα είναι ότι βρισκόμαστε σε επαφή με τις Ουγγρικές Αρχές και θα επανέλθουμε ενώπιον της Επιτροπής Αναφορών με μια αξιολόγηση όταν θα λάβουμε την απάντηση των Ουγγρικών Αρχών. Ευχαριστώ. Κυρία Γκόντς, σας ευχαριστώ. Άκουσα με χαρά μου ότι η Κομισιόν έρχεται σε επαφή με τις Ουγγρικές Αρχές, διότι εγώ θεωρώ ότι υπάρχει σημαντική πιθανότητα, διότι έχει αρχίσει μια αναθεώρηση της ε, φροντίδας πριν από τον τοκετό και ενδέχεται τελικά η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και ελπίζω μετά και η εφαρμογή της οδηγίας να γίνει σωστά. Διότι αυτό που βλέπουμε είναι, εγώ είμαι Ουγγαρέζα και είμαι και γιατρός. Γνωρίζω καλά λοιπόν την κατάσταση και είναι πραγματικά σοβαρή κατάσταση. η κατάσταση προκαλεί προβλήματα, όπως είπε και αναφερομένη. Για παράδειγμα, οι κεσαρικές τομές κατά αναλογία στην Ουγγαρία είναι πολύ, ε, πολύ ε, συχνότερες από ό,τι συνιστά ο ίδιος Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και από ό,τι είναι σε άλλες χώρες. Υπάρχει λοιπόν μια ε, στάση παρεμβατισμού η οποία καθαρά έχει σχέση με το οικονομικό και αναγκάζουν τις γυναίκες να εισάγονται στα νοσοκομεία για να γεννήσουν και όχι στο σπίτι σε οποιαδήποτε περίπτωση όπως είπα για λόγους οικονομικούς. Εφόσον μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο σωστά η οδηγία και δώσει έτσι και την ευκαιρία στο επάγγελμα της ΜΕΑΣ να αναπτυχθεί και να υπάρξει και, η απαραίτη, και, το απαραίτητο σώμα διατάξεων, ελπίζω ότι θα εξανθρωπίσει με τον τρόπο αυτό και την φροντίδα πρώτου το κοιτού και μετά από αυτόν. Πρέπει λοιπόν να παρακολουθήσουμε και την νομοθετική διαδικασία αλλά και την εφαρμογή της συγκεκριμένη οδηγίας στην Ουγγαρία και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει τον τομέα του το και του. Είναι στο τέλος της γραφής και θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων. Προτείνω και εγώ λοιπόν να διατηρηθεί ανοιχτή η αναφορά, αλλά παρακαλώ επίσης την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει, να έρθει σε επαφή με τις αρχές και με αυτή την έννοια, όχι μόνο για τα προσόντα δηλαδή. Ευχαριστώ κυρία Γκόντς, κυρία Άουκεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν είμαι ιατρός. Τίποτα από όλα αυτά. Και όταν άκουσα αυτά που είπε η κυρία από την Ουγγαρία νόμιζα ότι η κατάσταση είναι όπως ήταν στην Δανία πριν 44 χρόνια αλλά σε χειρότερη κατάσταση ήμασταν εντελώς ουδέτεροι απέναντι στα δικαιώματα των γυναικών, δεν υπήρχε ιατρική κάλυψη, αλλά υπήρχε βέβαια δυνατότητα επιλογής. Uh, ε, ο τοκετός δεν είναι ασθένεια, δεν πρέπει να την τοπίζουμε σαν μία ασθένεια, αλλά στο παρελθόν δυστυχώς αυτό ε, γινόταν και σε ορισμένες χώρες εξακολουθεί να γίνεται ακόμα. Σας ευχαριστώ λοιπόν κύριε Γκόντς για αυτά που είπατε. Άκουσα ότι το πρόβλημα δεν ισχύει μόνο για την Ουγγαρία. Υπάρχουν και άλλες χώρες όπου ισχύει αυτή η αντίληψη. Στη Λετωνία άκουσα ότι κάτι τέτοιο ισχύει, αλλά ότι άλλαξε ο νόμος πλέον και τώρα έχουν ελεύθερη επιλογή οι γυναίκες που θα γεννήσουν. Αν έχεις κάποια μέα να σε φροντίζει, σαν γυναίκα νιώθεις πραγματικά σε καλά χέρια. Θα πρέπει τα μέσα της δημόσιας υγείας να ασχολούνται με τα σοβαρά θέματα εκεί όπου πραγματικά τα χρειαζόμαστε. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ισχύει ένας τέτοιος νόμος. Γιατί δεν υπάρχει κάποιο οικονομικό συμφέρον καταρχάς το οποίο να εξυπηρετείται και να προτεύει. Αλλά τελικά κάποιος κερδίζει από αυτή τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος και στη συγκεκριμένη περίπτωση οι γιατροί. Και ε, το οικονομικά συμφέροντα των γιατρών είναι ένα θέμα, αλλά τα οικονομικά συμφέροντα της κοινωνίας είναι το βασικό θέμα. και πράγματι εφόσον υπάρχουν πραγματικοί επαγγελματίες με πραγματικά ε, επαγγελματικού επίπεδου τότε θα πρέπει να τις εμπιστευτούμε. Ευχαριστώ κύριος Μποστινάρο. Ε, και εγώ δεν είμαι γιατρός. Παρ' όλα αυτά έχω ορισμένες παρατηρήσεις να μου επιτρέψετε να κάνω, ξεκινώντας. να εμπνευστώ σε αυτά τα οποία θα πω από την κατάσταση στη χώρα μου και θα πρέπει να ανταλάβουμε υπόψη μας. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το θέμα αυτό σε επίπεδο κοινοτικό, σε επίπεδο ευρωπαϊκό σε ευρωπαϊκή κλίμακα, έτσι ώστε στα πλαίσια της εφαρμογής της οδηγίας και όχι απλά στους επιμέρους νόμους, να υπάρχει στο εσωτερικό της οδηγίας ένα πλαίσιο συνεκτικό για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος της ΜΕΑΣ. Αυτό αν γίνει ε, είναι κάτι που θα βοηθήσει και το επάγγελμα των ιατρών. Εφόσον υπάρχει ένα άλλο σώμα ε, επαγγελματικό, μια κατηγορία επαγγελματική, στη συγκεκριμένη περίπτωση οι που θα συνδράμουν τους ιατρούς. Να μην ξεχνάμε ότι τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας βρίσκονται σε βαθύτατη κρίση και αυτό προϋποθέτει ότι πρέπει να υπάρξει καλύτερη δαπάνη των διαθεσίμων πιστώσεων. Ταυτόχρονα επίσης ε, το μήνυμα το οποίο αποστέλω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι συνειδητοποιώντας ότι το επάγγελμα των, μεών αντιμετωπίζει τεράστιες ε, πιέσεις θα, από ένα τμήμα του, το, σώματος των ιατρών ε, που θέλουν να κάνουν επιχειρηματική δραστηριότητα εις βάρος των εγγύων και στα πλαίσια των τοκετών. Η τοκετή σαν παράδειγμα στις ιδιωτικές κλινικές είναι μια πανάκριβη διαδικασία, αλλά ακόμα και στα δημόσια νοσοκομεία που στην ουσία πολλές φορές παραπέμπουν τους ασθενείς τους απευθείας τους ιδιώτες ιατρούς. Θα πρέπει λοιπόν να διατηρηθεί το πλαίσιο λειτουργίας και δραστηριοποίησης ε, των μεών μια πιο συνεκτική και μια πιο ουσιαστική νομοθετική ρύθμιση σε κοινοτικό επίπεδο θα βοηθήσει και τις απομεμακρυσμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου η παρουσία των μεών είναι απαραίτητη και πολύτιμη και όπου μια κανονική διαδικασία το κετού μπορεί να μετατραπεί σε μια κατεπίγουσα διαδικασία όπου η ιατρική παρουσία θα είναι απαραίτητη και δεν είναι δυστυχώς πάντα διαθέσιμη. Λοιπόν, πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει το θέμα σφαιρικά και να προχωρήσει σε έναν διαφθρωτικό διάλογο με τα κράτη-μέλη και με τα εθνικά συστήματα για να λειτουργήσει το σύστημα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο προς όφελος όλων και να πιέσει την Ουγγρική κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματα των αναφερόντων. Γιατί πράγματι από τις θέσεις που εξέφρασαν οι αναφέροντες οι ε, γυναίκες έχουν να κερδίσουν και δεν πρέπει οι ιδιωτικές κλινικές να ελέγχουν τα πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος το λόγο. Ένα λεπτό έχετε να απαντήσετε, ε, αναφέρετε στην αναφερόμενη πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ακούσαμε πάρα πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά τα σχόλια. Θα ήθελα να προσκαλέσω την Επιτροπή Αναφορών να εξετάσει ε, προσεκτικά την πρόταση νόμου την οποία αυτή τη στιγμή κατέθεσε η Ουγγρική κυβέρνηση και που θεωρώ ότι δεν είναι συμβατή η νομική αυτή ρύθμιση με την οδηγία. Από την άλλη τίθεται και το θέμα της πρακτικής εφαρμογής αυτών των νομικών ρυθμίσεων. Ελπίζω να μπορέσουμε, αν θέλετε, ακόμα περισσότερες πληροφορίες να σας δώσουμε για να πάρετε τις σωστές αποφάσεις ευχαριστώ που μας φέρατε την περίπτωση αυτή ε, στην επικαιρότητα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κρατήσει την αναφορά ανοιχτή. Ελπίζω να μην χρειαστεί πάρα πολλής χρόνος έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ολοκληρώσει ε, την προσπάθεια την οποία κάνει και να συναντηθούμε για να δούμε σε ποιο σημείο θα έχουμε φτάσει. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, την 1380 του 2011 από τον Ούγκρο πολίτη κύριο Τάκ για την Εταιρεία Προστασίας της Ανατολικής Ουγγαρίας σχετικό με την προστασία της πανίδας και της χλωρίδας γύρω από την πόλη Γκιόρ της Ουγγαρίας. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Τάκ. Ευχαριστώ πολύ. Απευθύνομαι στην Επιτροπή Αναφορών. Κυρία Πρόεδρε, στις 24 Ιανουαρίου του 2011, μέσω της αποφάσεώς σας, ζητήσατε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στραφεί προς την περίπτωση της ε, Ουγγαρίας, κυρίως όσον αφορά την επέκταση μιας αυτοκινητοβιομηχανίας έξω από την πόλη Γκιόρ της ε, Ουγγαρίας. Ε, πρόκειται για επέκταση της αυτοκινητοβιομηχανίας σε μία περιοχή η οποία έχει ιδιαίτερα πλούσια αλλά και προστατευόμενη χλωρίδα και πανίδα. Στα πλαίσια της περιοχής αυτής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δαπανίσει πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ ε, για το πρόγραμμα LIFE το 2009. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε τα σχέδια επέκτασης αυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας. Μέχρι τώρα δε δεν έχει δώσει ρητά και επίσημα την σύμφωνη γνώμη της για την επέκταση της εν λόγω αυτοκινητοβιομηχανίας σε αυτήν την ε, περιοχή η οποία προστατεύεται από το πρόγραμμα LIFE η αυτοκινητοβιομηχανία αλλά και η ουργική κυβέρνηση διατείνονται ότι έχουν όλες τις απαραίτητες θετικές γνωμοδοτήσεις Ωστόσο, δεν έχουμε εμείς λάβει γνώση αυτών των ρητών συμφώνων αποφάσεων. Σαφώς αναφέρεται ότι ε, ε, στην αντίστοιχη περίπτωση της Πορτογαλίας είχε επιτραπεί ε, η οικοδόμηση της ε, αντίστοιχης ε, βιομηχανίας, γιατί εκεί δεν υπήρχε καμία εναλλακτική λύση. Στην προκείμενη περίπτωση όμως της Ουγγρικής πόλεως Γκιόρ ε, υπάρχουν δυνατότητες εναλλακτικής επίλυσης του προβλήματος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα, μια άλλη έκταση στην πόλη της Ζίξορ και όχι στην πόλη Γκιόρ. Ε, πρόκειται για ε, πόλη η οποία βρίσκεται πιο μακριά από την περιοχή Life. Πρόκειται για ε, λιγότερο κατοικημένη και με μικρότερο πληθυσμό πόλη και επομένως αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει μια ορθή εναλλακτική λύση, μια βιώσιμη εναλλακτική λύση. Επίσης, μη λησμονούμε ότι υπάρχει ήδη μια ε, αυτοκινητοβιομηχανία σε, κοντινές, ε, σε κοντινή περιοχή και θα μπορούσε να μεγαλώσει εκείνη η εγκατάσταση. Οι ε, Ουγγρικές αρχές πρέπει να πούμε ότι έχουν υποσχεθεί αντισταθμιστικά μέτρα για την ενδεχόμενη ζημία η οποία θα προκληθεί στο περιβάλλον. Ωστόσο πρόκειται για οικονομική αντισταθμιστικά ε, μέτρα τα οποία φυσικά δεν λαμβάνουν υπόψη την πραγματική προστασία του περιβάλλοντος. Επομένως, τα όσα μέτρα περιβαλλοντική κακής ε, αντιστάθμισης αναφέρονται, φρονούμε πως δεν είναι ικανοποιητικά και ικανά. Ε, πρόκειται εδώ για περιοχές οι οποίες καλύπτονται από την ε, Natura, από το πρόγραμμα Natura 2000 και επομένως μιλάμε για ιδιαίτερα ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές. Στην περίπτωση της Ουγγαρίας έχουμε ε, ένα, ε, μια περιοχή Natura ε, η οποία είναι εξαιρετικά μεγάλη και πολύ μεγαλύτερη μάλιστα από την αντίστοιχη περίπτωση ε, του αεροδρομίου ε, ε, του Λούμπεκ. Και ωστόσο τα αντισταθμιστικά μέτρα τα οποία προτείνονται εδώ είναι ίδια με αυτά που είχαν προταθεί για το αεροδρόμιο Λούμπεκ. Η Κομισιόν θα πρέπει οπωσδήποτε να μελετήσει τα αντισταθμιστικά μέτρα τα οποία προτείνονται σε εθνικό επίπεδο. Οι εθνικές ουγγρικές αρχές διατείνονται ότι η Κομισιόν έχει μελετήσει και έχει δώσει πράσινο φως για αυτό το σύστημα αντισταθμιστικών ε, μέτρων. Ε, όμως εμείς δεν έχουμε στοιχεία ότι έχει ληφθεί όντως αυτή η απόφαση ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρόλα αυτά, ε, η, η ίδια η επέκταση, το σχέδιο αυτό της επέκτασης έχει ήδη ε, εγκριθεί. Ε, πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να συζητηθεί το ζήτημα αυτό. Μάλιστα, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής στην απόφαση του της 13ης Μαρτίου του 2012 είχε αποφανθεί ότι καμία συγκεκριμένη απόφαση απόφαση ε, δεν είχε ε, ε, και απάντηση δεν είχε δοθεί στον αναφέροντα. Στις τρεις εβδομάδες οι οποίες ακολούθησαν την απόφαση παράτασης επίσης δεν απεστάλησαν οποιασδήποτε αποφάσεις οι πληροφορίες τις οποίες είχαμε ζητήσει δεν παρελήφθησαν ποτέ. Πληροφορίες οι οποίες θα είχαν ε, μπορέσει να χρησιμοποιηθούν για να ενισχυθεί ο φάκελος ε, της ε, αναφοράς μας. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, Δεχόμαστε βεβαίως ότι η στρατηγική για την βιοπικιλότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να γίνει σεβαστή και όντως το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θέλει να στηρίξει οπωσδήποτε κάποια βιομηχανική πρόοδο και κάποια προγράμματα τα οποία αποσκοπούν στη βιομηχανική πρόοδο, όμως ε, αυτό δεν θα πρέπει να γίνει με ζημία και καταστροφή προστατευόμενων οικοσυστημάτων. Πρόκειται ε, για στοιχεία τα οποία ε, ε, στην ουσία παραπέμπουν στην καταστροφή του, του Αμαζονίου και των τροπικών δασών. Ευχαριστώ πολύ. Uh, yes, thank you, madam. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πράγματι, τον Ιανουάριο του 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μια θετική άποψη για το αναπτυξιακό σχέδιο του Γκιόρ, το οποίο υπέβαλαν οι Ουγγρικές αρχές. Να θυμίσω εδώ λίγο το πλαίσιο στο οποίο έγινε αυτό. Η οδηγία αποκλείει ε, την δυνατότητα βλάβης στις περιοχές Natura 2000, όμως υπάρχουν ορισμένες προβλέψεις οι οποίες δίνουν την δυνατότητα για εξαιρέσεις και οι εξαιρέσεις αυτές θα πρέπει ε, να ε, εκπληρούν ορισμένες προϋποθέσεις. Πρώτον, να υπάρξει μια ουσιαστική μελέτη επιπτώσεων. Δεύτερον, να υπάρξει απόδειξη για την έλλειψη εναλλακτικών περιοχών. Ε, να ονομα, να, να δοθούν στην, ε, ε, στην, ε, στο κοινό οι λόγοι για τους οποίους δεν μπορεί να γίνει σεβαστό το κοινό συμφέρον στην συγκεκριμένη περίπτωση και αφού πήρε τα στοιχεία αυτά από την Ουγγρική κυβέρνηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο ότι οι προϋποθέσεις αυτές σχετικά με το σχέδιο το χωροτακτικό του Τζερ έγιναν δεκτές. Έκαναν την ανάλυση των εναλλακτικών λύσεων, κατέληξαν στην εξέταση κάποιων εναλλακτικών προτάσεων σε ευρύτερο εδαφικό πλαίσιο στην Ουγγαρία γύρω από την πόλη του Τζερ και κατέληξαν στο ότι καμία από τις υπόλοιπες εναλλακτικές προτάσεις δεν ήταν κάτι το εφικτό λόγω συγκεκριμένων κριτηρίων και ελλείψεων όπως το μέγεθος της έκτασης, έλλειψη συγκοινωνιακών υποδομών κτλ. Σχετικά με τους λόγους μη σεβασμού ε, του ε, κρατικού συμφέροντος, οι Ουγγρικές αρχές έδωσαν ορισμένες πιστικές εξηγήσεις ότι η επέκταση αυτή θα δημιουργήσει άμεσα και έμεσα αρκετές χιλιάδες θέσεις απασχόλησης και σε επίπεδο αντισταθμιστικών μέτρων Γενικά θα αναπτυξιακά θα βοηθηθεί πολύ η περιοχή και η συγκεκριμένη πόλη και γι' αυτό εξέδωσε θετική άποψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η γνωμοδότηση αυτή βέβαια δεν προκαταλαμβάνει την εσωτερική εθνική διαδικασία αδειοποίησης στην Ουγγαρία. Οι Ούγγροι θα ολοκληρώσουν την διαδικασία αυτή από μόνοι τους όταν το κάνουν. Συνεπώς ο αναφερόμενος ήρθε ο αναφέρον συγγνώμη, ήρθε σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με νέα επιχειρήματα διαφωνώντας με την τεκμηρίωση της Ουγγρικής κυβέρνησης. Εμείς απαντήσαμε στο νέο αίτημα αναθεώρησης ε, του, του αναφέροντος διαφωνώντας μαζί του και συμφωνώντας με τις αρχές. και ε, μετά υπέβαλε νέο αίτημα στην Επιτροπή σας ο αναφέρον και εμένουμε σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η αναπτυξιακή αυτή δράση ήταν συμβατή με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ η κυρία Άουκεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εδώ και κάποια χρόνια είχαμε διατυπώσει μια έκθεση στο εσωτερικό της έκθεσής μας η οποία έλεγε, αναφερόταν μάλλον, στον τρόπο με τον οποίο ε, η οδηγία Natura 2000 γίνεται σεβαστή ή όχι. Ένα από τα συμπεράσματα στα οποία είχαμε καταλήξει ήταν ε, ότι δεν υπήρχε σωστή ανάλυση των εναλλακτικών προτάσεων. Πάντα είχαμε την τάση να λέμε ότι εφόσον η κυβέρνηση και η κεντρική διοίκηση λέγει ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, ε, so be δεν υπήρχε άλλη λύση. Έτσι λοιπόν τώρα βλέπουμε ότι ναι μεν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι έχει υπάρξει μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την οποία όμως εμείς δεν έχουμε στη διάθεσή μας. Εφόσον έχει υπάρξει μια τέτοια ανάλυση, η οποία πράγματι αποδεικνύει ότι οι εναλλακτικές προτάσεις δεν ήταν εύκριστες για κάποιους λόγους, να το δούμε. Αν είναι πιο εύκολο ε, και λιγότερο ε, και περισσότερο ευθυνό να χρησιμοποιηθούν τέτοιες περιοχές να γίνει αυτό, αλλά πρέπει όμως να έχουμε αποδείξεις εδώ λίγο, γιατί μου έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι το κράτος της Ουγγαρίας στη συγκεκριμένη περίπτωση το μόνο που λέει είναι κοιτάξτε εμάς μας ενδιαφέρει να δημιουργηθεί μια μονάδα η οποία θα ανοίξει θέσεις εργασίας. Όλα τα άλλα δεν μας ενδιαφέρει. και όπως είχε πει και ο Μπαρόσο, ο σεβασμός της Natura 2000 είναι σημαντικός, αλλά όταν έχει τη δυνατότητα να το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα το κάνει. Και φοβάμαι ότι αυτή η απαράδεκτη στάση χαρακτηρίζει και την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ λοιπόν προσωπικά θα ήθελα να έχω στην διάθεσή μου παρακαλώ την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα ήθελα επίσης ε, να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα λεγόμενα ε, αντισταθμιστικά ωφέλη. Θα ήθελα να έχω περισσότερα στοιχεία και να μας πούν και οι αναφέροντες εάν πράγματι ε, είναι τρόπο τον οποίο έπρεπε μαζί τους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή μήπως θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρενέβη έτσι ώστε να δημιουργήσει, να λειτουργήσει σαν τροχοπέδι στις διαδικασίες των πολιτών της Ουγγαρίας γιατί έχουν υπάρξει και τέτοιες περιπτώσεις. θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα να ζητήσουμε και από την διαμεσολαβήτρια να μας πει αν είναι ικανοποιημένη από τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τους αναφέροντες. Εμείς προσπαθούμε να είμαστε δραστήριοι υπέρ των πολιτών. Για να το κάνουμε αυτό όμως πρέπει να έχουμε τα απαιτούμενα μέσα, γνώση, στοιχεία στη διάθεσή μας. Αν τα έχουμε εγώ δεν το έχω πάρει είδηση. Συνεπώς η εντύπωσή μου είναι ότι από ουγγρικής πλευράς επιλέγει επελέγει η φθηνότερη λύση και όλα τα άλλα είναι λεπτομέρειες. Όχι, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση μάλιστα υπάρχουν και κοινοτικά κονδύλια τα οποία χρησιμοποιούνται για την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν μ' αρέσει αυτή η υπόθεση. Θυμίζω την πολωνική περίπτωση αντίστοιχη την οποία είχαμε αντιμετωπίσει και εκεί καταφέραμε νομίζω μια νίκη περηφανή για την προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ούκεν, λέει η Πρόεδρος. Παρακαλώ. Θα ήθελα να πω και εγώ δύο λόγια. Είμαι αρχιτέκτονας και από επαγγελματική απόψεως πρέπει να πω ότι θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ε, αυτούς που θα κατοικήσουν την περιοχή που κατοικούν ήδη. Διότι ε, ε, κάποιοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, αξιωματούχοι οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις αυτές που ζουν όμως χιλιόμετρα, χιλιάδες χιλιόμετρα ή εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά ε, δεν μπορούμε να τους λάβουμε υπόψη μας, δεν καταλαβαίνουν τι υποφέρουν, ε, πόσο υποφέρουν οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν δίπλα σε αυτές τις εγκαταστάσεις. Αυτοί θα πρέπει να γνωμοδοτήσουν και η γνώμη αυτών των ανθρώπων που ζουν εκεί κοντά θα πρέπει να να ληφθεί υπόψη. Αυτοί οι οποίοι μένουν χιλιάδε χιλιόμετρα μακριά είτε στι Βρυξέλλες είτε στην πρωτεύουσα της Ουγγαρία. προφανώς δεν είναι σε θέση να καταλάβουν το μέγεθος του προβλήματος. Ευχαριστώ. Πρόεδρο. ευχαριστούμε πολύ. Ένα λεπτό έχετε στη διάθεσή σας ε, για να απαντήσετε κατόπιν όσων ακούσατε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε λέει ο κύριος Ζακ, θα ήθελα να πω τα εξής. Στα πλαίσια της ε, διαδικασίας που μας απασχολεί δεν υπήρξε καμία επίσημη ακρόαση. Ε, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2011 διοργανώθηκε μια διαδικασία διαβούλευσης με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών ε, χωρίς στήριση πρακτικών, επομένως με τελείως ανεπίσημο τρόπο. Επίσης, στις Βρυξέλλες όταν οργανώθηκε ε, μια πιο επίσημη συνάντηση, εμείς δεν είχαμε καν προσκληθεί και επομένως δεν είμαστε καθόλου σε θέση σαν εκπρόσωποι των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ε, να είμαστε παρόντες και να πάρουμε μέρος σε αυτήν την πιο επίσημη διαβούλευση. Ε, πάντα μας είπαν ότι δεν μπορούσε να γίνει τίποτα, ότι δεν μπορούσε να αλλάξει καμία απόφαση ε, και ότι στο μέλλον θα έγινε το κάποια προσπάθεια αντιστάθμισης κτλ σε καμία περίπτωση οι δικές μας ε, παρατηρήσεις ε, δεν ακούστηκαν και οπωσδήποτε οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών δεν είχαν σε καμία ε, περίπτωση και σε καμία χρονική στιγμή την δυνατότητα να υποβάλουν τις εναλλακτικέ λύσεις οι οποίες είχαν προκύψει μετά από συναντήσεις με εμπειρογνώμονες. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, δεν νομίζω ότι από τις πληροφορίες που έχουμε ε, λάβει μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχει κλείσει το θέμα όσον αφορά την ε, ε, περί λόγος αναφορά. Ε, επίσης και όπως υπογράμμισε και η Σόκεν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη και ανάλογες περιπτώσεις στις οποίες η αντίδρασή της ήταν διαφορετική. Θα πρέπει να μελετήσει περαιτέρω λοιπόν ε, την αναφορά αυτή η οποία βασίζεται σε πάρα πολύ ε, συγκεκριμένη τεκμηρίωση την οποία έχει υποβάλει ο αναφέρον. Έχουμε ήδη μια γνωμοδότηση επί του σημείου αυτού, αλλά καλό θα ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη το αίτημα του κυρίου Ζακ ε, και να μελετηθεί η αναφορά αυτή και από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Εγώ λοιπόν προτείνω ε, να αφήσουμε ανοιχτή το το αίτημα αυτό. Να αφήσουμε λοιπόν την αναφορά ανοιχτή τεκμέρο δε και από τις παρεμβάσεις των συναδέλφων ότι συμφωνούν ε, απολύτως. Να μελετηθεί περαιτέρω λοιπόν ε, ε, ό,τι σχετίζεται με την εν λόγω αναφορά να σταλεί και η τεκμηρίωση σε την Επιτροπή Περιβάλλοντος έτσι ώστε να γνωμοδοτήσει και η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Αυτά είχαμε να πούμε λοιπόν για τούτη την αναφορά για σήμερα. Ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά τον κύριο Ζάκ και περνούμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως. Είναι το ε, σημείο υπεριθμών 10, αναφορά 1342 κάθετος 2011 ε, που έχει υποβάλει η κυρία Γκραματσκή, γερμανικής ηθαγένειας, εκ μέρους της οργάνωσης ορθινολογίας Μαύρος Πελαργός, σχετικά με την παράβαση της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, της οδηγίας περί περιβαλλοντικής ευθύνης, καθώς και τη σύμβαση του Άρχους για την περιοχή Σαν Μπερναμπέ. Η κυρία Νοέλια Γιουράδο Ορτέγα θα πάρει το λόγο. Θα μας κάνει δε μία παρουσίαση σε PowerPoint. Για πέντε λεπτά έχετε το λόγο κυρία μου. Ε, bueno, es imposible explicar en cinco minutos. Είναι πάρα πολύ δύσκολο μέσα σε πέντε λεπτά να πει κανεί δέκα χρόνια προσπάθειας. Θα προσπαθήσω με ταχύτητα όμως να σας μεταφέρω αυτά τα οποία λέει. Μιλάμε για την περιοχή κοντά στο Αλχεσίρας απέναντι από το Γιβλαρτάρ. Ξέρετε πως υπάρχουν θέματα για τη διαχείριση της ε, περιοχής ανάμεσα. Είναι σταυροδρόμοι θα έλεγα μεταναστευτικών αποδημητικών πτηνών ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Αφρική. Έρχονται εκεί προλες φορές για να χρησιμοποιήσουν τους υδάτινους πόρους της περιοχής. Βλέπετε μια εναέρια εδώ άποψη της περιοχής Υπάρχει από τη δεκαετία του 80 μια επιφανειακή μεταλλευτική δραστηριότητα. Έχει δημιουργηθεί ένας χώρος δεύτερης επεξεργασίας, εξόριξης όπως ονομάζεται και έχει δημιουργηθεί μια νέα περιοχή υδροτόπου στο σημείο 2. Εδώ βλέπετε το τρίτο σημείο που είναι η, το, η κατεξοχήν περιοχή ε, των, ε, της ε, εξορρυκτικής εκμετάλλευσης. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε και κατασκευές πάνω σε προϊστορικά μνημεία αρχαιολογικής σημασίας. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα επίσης με την μόλυνση των υδάτινων πόρων και την παραβίαση των κοινοτικών νόμων. Βλέπουμε εδώ ότι ο κίνδυνος είναι σαφής για την μόλυνση των υδάτινων πόρων. Ξεκίνησε από τη δεκαετία του 80 Βλέπετε ότι έχουμε το σημείο 2 που δημιουργήθηκε ένας νέος υδρότοπος παραβιάζοντας την ισχύουσα οδηγία. Είχε υπάρξει ε, πριν ξεκινήσει η εξορεκτική διαδικασία μια δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά αυτό από τότε δεν έχει ελεγχθεί. και εδώ παραβιάζεται η οδηγία υπαριθμών 85 του 2007. Βλέπετε εδώ μία εικόνα δορυφορική, 5 Ιουλίου του 2003. Ξέρουμε ότι την ίδια περίπου εποχή είχε υπάρξει και η κατάθεση της περιβαλλοντικής μελέτης. Ήδη το 2008 δημιουργήθηκε μια, ένα σύλλογος, ο Φαπάξα, καταγγέλλοντας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα γεγονότα αυτά για πάρα πολλά χρόνια. Στην ουσία έχουμε να κάνουμε με ένα κρυφό σημείο απόρριψης των... Μια κοχωματερή, εν πάση περιπτώσει, ήδη από το Μάρτιο του 2011 δεν είχε απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις ερωτήσεις τις οποίες είχαμε εμείς θέσει. Ποιες είναι τώρα οι προθέσεις των Ισπανικών αρχών να καλύψουν τον υδρότοπο αλλά έχει σταματήσει η διαδικασία αυτή λόγω της αντίδρασης των τοπικών συλλόγων και οργανώσεων Υπήρξαν καταγγελίες και προς τον Ισπανό διαμεσολαβητή. Έχουμε επίσης φτάσει και στην εισαγγελική αρχή για την προστασία του περιβάλλοντος του Αλχεσίρας, όπου δυστυχώς το αίτημά μας στέθηκε στα αρχεία. Και αυτό μας έδωσε να καταλάβουμε ότι η αρμόδια εισαγγελική αρχή Una administración pasa la pelota a otra, a otra administración, quienes a su vez cambian continuamente. Ε, βλέπουμε εντωμεταξύ ότι η επιχείρηση αυτή αλλάζει συνεχώς όνομα και αυτό δημιουργεί τυπικά προβλήματα στους τρόπους με τους οποίους οι τοπικές αρχές αντιμετωπίζουν το θέμα και δεν γίνεται έτσι σεβαστή η συνθήκη του άρχους. Και από το 2013 η εταιρεία έχει κάνει μια δήλωση ε, για την τροποποίηση της περιβαλλοντικής μελέτης του 2003. Παρ' όλα αυτά έχει καταλήξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο συμπέρασμα ότι δεν έχει υπάρξει ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής και δυστυχώς θα έχει πεθάνει το περιβάλλον όταν αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει το θέμα. Δεν υπάρχει ποιότητα στην περιοχή, έλεγχος της ποιότητας των δραστηριοτήτων έχουν κοπεί πάρα πολλά δέντρα τα οποία ήταν ηθαγενή της περιοχές ε, και δεν έχουν ξαναφυτευτεί εκ νέου. Έχει μολυνθεί το νερό, ε, η υδάτινη πόρη. Δεν έχει γίνει σεβαστή η οδηγία του 2035 του 2004 και δεν έχει εφαρμοστεί η διαδικασία που αφορά το Natura 2000. Ε, Παρ' όλα αυτά και τα πουλιά και οι κάτοικοι της περιοχής, τα αποδημητικά πουλιά έχουν ανάγκη από καθαρό νερό ε, για ε, την δική τους κατανάλωση, για την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα. Εμείς θα θέλαμε να να προσπαθήσετε να κάνετε μία επίσκεψη στην περιοχή μας. γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος από τα διάφορα μέταλλα τα οποία έχουν απορριφθεί. Υπάρχουν παραδείγματα από χώρες όπως η Γερμανία, η Αγγλία και η Αυστρία. Σας ευχαριστώ. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν ξέρω, θα πρέπει να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Χωσεμαρία Ράμος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πράγματι, η συγκεκριμένη αναφορά, όπως είπες και ο αναφέρον, αφορά την εξορεκτική δραστηριότητα στην περιοχή του Σαν Μπερναμπέ, στην αυτόνομη περιοχή της Ανδαλουσίας, στο Καδί της Ισπανίας. Ο αναφέρον καταγγέλει τις βλάβες που έχει, το που έχει υποστεί το περιβάλλον από τη δραστηριότητα αυτής της εξορεκτικής δραστηριότητας μετά από τις άδειες τις οποίες εξέδωσαν οι τοπικές αρχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε υπόψη της λοιπόν το θέμα μετά από μια κοινοβουλευτική ερώτηση και με την συγκεκριμένη αναφορά η οποία κατατέθηκε το 2011 και γι' αυτό ξεκίνησε μια ερευνητική διαδικασία μέσω του μηχανισμού EU Pilot, το οποίο χρησιμοποιείται για να τεθούν ερωτηματικά προς τα κράτη-μέλη και απευθύνθηκε επανειλημμένα προς τις Ισπανικές αρχές ζητώντας τις παρατηρήσεις του σχετικά με τις καταγγελίες του αναφέροντος και σχετικά με τον σεβασμό της κοινοτική νομοθεσίας που αφορά το περιβάλλον στη συγκεκριμένη περιοχή. Ο θεματοφύλακα της συνθήκης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ελέγξει την, τον σεβασμό ε, του κοινοτικού δικαίου, έχει την δυνατότητα να ερευνήσει λοιπόν ε, την διαδικασία αυτή επί τη βάση των αποδείξεων και των τεκμηρίων που καταθέτει και ο αναφέρον, όπως επίσης και των στοιχείων τις οποίες, τα οποία αποστέλουν οι αρμόδιες τοπικές αρχές. Εμείς πήραμε εκθέσεις και από την περιφερειακή αυτόνομη περιοχή και από την κυβέρνηση την τοπική και από τις αρμόδιες αρχές για την προστασία του περιβάλλοντος. Θα πρέπει στα πλαίσια λοιπόν της διαδικασίας σεβασμού της κοινοτικής νομοθεσίας. Υπήρξε μία στο παρελθόν μελέτη ε, ε, επιπτώσεων στο περιβάλλον τον Ιούνιο του 2003 που ενεκρίθη από την Περιφερειακή Αρχή του Καδίζ στην Ισπανία, στην Ανδαλουσία. Η, ε, η συγκεκριμένη μελέτη επιπτώσεων δημοσιεύθηκε στην αρμόδια επίσημη εφημερίδα στο επίσημο δελτίο του Καντίζ στα τέλη του 2003 σχετικά με την ε, οδηγία 85 του 2003 η οποία οδήγησε στο τελικό κείμενο της ε, οδηγίας του 2011 που συγκεντρώνει το σύνολο των ρυθμίσεων που υπήρχαν μέχρι τότε. Δόθηκε η άδεια λοιπόν για την εκμετάλλευση αυτού του ανοιχτού λατομείου η οποία τερματίστηκε το 2011 και η μοναδική δραστηριότητα η οποία επιτρέπεται πλέον είναι το σχέδιο αποκατάστασης ε, που προέβλεπε η διαδικασία της κατάθεσης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων το 2003 και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αναλάβει η συγκεκριμένη εξορεκτική ε, επιχείρηση την αποκατάσταση του εδάφους και της περιοχής. Υπάρχουν οι διάφορες κοινοτικές οδηγίες όπως η οδηγία για τους οικοτόπους και η Natura 2000 Ε, έχει υπάρξει μια μακρά περίοδο συζήτησης και ρυθμίσεων εναντίον της ε, ε, Ισπανίας έτσι ώστε να καθορίσει σωστά τις περιοχές Natura 2000. Το 25% περίπου του εδάφους της Ισπανικής επικράτειας περιλαμβάνονται στο Natura 2000. Απευθυνθήκαμε στις αρμόδιες αρχές και ε, φαίνεται ότι οι εξορυκτικές αυτές δραστηριότητες σε καμία περίπτωση δεν σεβάστηκαν τους απαραίτητους κανόνες και δεν συμπεριελήφθη η περιοχή στις περιοχές οι οποίες ελέγχονται από τις ρυθμίσεις των περιοχών Natura 2000. Από νομικής επόψεως αυτή, αυτός ο τεχνητός ε, υδρότοπος ο οποίος δημιουργήθηκε ε, παραβιάζει γενικά πολλές ρυθμίσεις και ταυτόχρονα όμως δεν την χάνει ειδική προστασία όπως οι περιοχές οι οποίες περιλαμβάνονται στη Natura 2000. Οι τοπικές αρχές και στη συγκεκριμένη περίπτωση η ε, Δημοτική Αρχή του Αλχεσίρας ανέφεραν διαδικασίες οι οποίες ξεκίνησαν εναντίον της επιχείρησης για τη μη εκπλήρωση των ανηλυμένων της υποχρεώσεων. Οι Ισπανικές αρχές μας ενημέρωσαν επίσης ότι η εισαγγελία περιβάλλοντος που έχει εκτελεστικές εξουσίες επί της συγκεκριμένης περιπτώσεως έχει ξεκινήσει διαδικασίες τις οποίες έφερε εις γνώση μας. Οι υπηρεσίες λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέλησαν την περίπτωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως θέμασοφύλαξη της συνθήκης αυτό το οποίο μπορεί να κάνει είναι να συνεργαστεί και να ζητήσει από τις τοπικές αρχές τον σεβασμό των κοινοτικών αρχών τον σεβασμό της κοινοτικής νομοθεσίας. Αλλά δεν μπορούμε να στραφούμε εμείς εναντίον της συγκεκριμένης επιχείρησης, πρέπει οι τοπικές αρχές να το κάνουν αυτό. Συμπερασματικά λοιπόν και αφού εξετάσαμε το σύνολο των στοιχείων τα οποία είχαμε στη διάθεσή μας, δεν μπορούμε εμείς να καταλήξουμε σε μία παραβίωση του κοινοτικού δικαίου. Ευχαριστούμε τον αναφέροντα για τα στοιχεία τα επιπλέον τα οποία μας έδωσε σήμερα και θα καταλήξω λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τις αρμόδιες ισπανικές αρχές να μας ενημερώσει για την κατάληξη της διαδικασίας αυτής και των κυρωτικών διαδικασιών οι οποίες έχουν ξεκινήσει εις βάρος της επιχείρησης. Μου έχετε ζητήσει εσείς τώρα το λόγο. Ο κύριος Φερνάντες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον αναφέροντα, την αναφέρουσα μάλλον, Υπάρχουν διάφορα θέματα στα οποία θα ήθελα να σταθώ εδώ και θα ήθελα να διευκρινίσουμε κάποια θέματα. Ε, στρέφομαι προς τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πράγματι γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει δικές της ερευνητικές ε, ε, δυνατότητες και εξαρτάται ως προς αυτό από τις αρμόδιες τοπικές αρχές παρόλα αυτά έχει λάβει υπόψη της και τις ισχύουσες ε, ρυθμίσεις νομοθετικές για την προστασία του περιβάλλοντος και τον τρόπο που εφαρμόζονται από τις τοπικές αρχές. Το θέμα είναι αν προχωράει ικανοποιητικά έτσι και αλλιώς και το σχέδιο αποκατάστασης των περιοχών αυτών. Δεν έχω στοιχεία από αυτό. Θα σας δώσω το λόγο στο τέλος της διαδικασίας. Θα μπορέσετε να πάρετε τελευταία το λόγο. Πρώτα θα μιλήσουν οι διάφοροι συνάδελφοι. Ε, αν θέσουν ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν ξέρω αν τελειώσατε κύριε Φερνάντες. Νομίζω ότι από τα στοιχεία τα οποία μας έδωσαν οι αναφέροντες ε, και στο παρελθόν η κατάσταση παρουσιάζεται με πάρα πολύ περίεργο τρόπο. Εφόσον αυτό το άγνωστο ε, για τους αναφέροντες σε σχέδιο αποκατάστασης της περιοχής ε, αποκαθιστά τις ζημίες ε, τις οποίες, οι οποίες έχουν υπάρξει όπως η μόλυνση σαν παράδειγμα των υδάτινων πόρων και μπορούν να δημιουργήσουν ένα υδρότοπο ο οποίος να εξυπηρετεί γενικά τα αποδημητικά τα οποία περνούν από εκεί στο μέλλον να αποκαταστήσει εν πάση περιπτώσει στην φύση, στην περιοχή και το περιβάλλον της περιοχής. Να πω επίσης ότι σχετικά με τις πληροφορίες που έστειλε η κυβέρνηση η τοπική προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν ήταν αηφόρος η επένδυση αυτή από ό,τι φαίνεται βραχή πρόθεσμα ε, Θα ήθελα να μάθω αν άλλα αντίστοιχα στοιχεία τα οποία έστειλε η συγκεκριμένη τοπική κυβέρνηση σε επίπεδο τεχνικό και τα λοιπά ήταν πράγματι ικανοποιητικά. Γιατί μερικές φορές τέτοιου είδους διοικήσεις έρχομαι από την Ισπανία και γνωρίζω δεν είναι ικανοποιητικές. Θα ήθελα να παραμείνει ανοιχτή η διαδικασία λοιπόν αυτή και να ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίως από τις τοπικές αρχές και ιδιαίτερα από την περιφερειακή κυβέρνηση όπως και από τους δημοτικούς άρχοντες του Αλχεσίρας. Κύριε Μποστινάρου, πάρα πολύ γρήγορα γιατί έχουμε καθυστερήσει. Ναι, λοιπόν, πολύ σύντομα. Πρώτο, η Κομισιόν αναφέρθηκε μόνο στη μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου. Σωστό αλλά εγώ θα ήθελα να λάβει η Κομισιόν υπόψη και την ήδη τροποποιημένη από το Κοινοβούλιο οδηγία για την μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου και τα νέα στοιχεία τα οποία θα ε, διαπούν και, τους, ε, και τις νέες ρυθμίσεις, δηλαδή την ουδετερότητα και την κειμενικότητα του εκτιμητού. Επίσης την υποχρεωτική συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών, stakeholder, δηλαδή κοινή γνώμη, ε, μη κρατικών οργανισμών κλπ. Είτε ατομικά είτε με τρόπο οργανωμένο. Τρίτο, πού βρίσκεται λοιπόν εδώ, σε αυτά που λέτε η αρχή του ορυπαίνων πληρώνει. Για να αποκαταστήσουν το τοπίο, ναι, να, το αποκαταστήσουν το τοπίο, αλλά όχι όπως θέλουν με αυθαίρετο τρόπο. Υπάρχουν ξεκάθαρες προβλέψεις και υποχρεώσεις που απορρέουν από την μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου που γίνεται στην αρχή της διαδικασίας. Ο μόνος τρόπος που μπορεί να γίνει είναι να εφαρμόσουν σωστά τα όσα ρητά περιλαμβάνει η μελέτη αντικτύπου. Εγώ θέλω να δω αυτή την αξιολόγηση που δεν τη βλέπω. Τέλος, με συγχωρείτε που βήχω, είναι γεγονός ότι δεν μπορεί κανείς να επαφίεται μοναχά σε μονόπλευρες πληροφορίες, ανεξαρτήτως του ποια είναι η πλευρά αυτή, είτε δηλαδή είναι η αναφερόμενη, είτε είναι η εταιρεία ή οι αρχές. Είναι χρέος σας να ψάξετε, να ελέγξετε και να ξαναελέγξετε, ώστε να είστε βέβαιοι ότι η μελέτη αντικτύπου, η αξιολόγηση διαδικασίας δηλαδή, ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι αν παραμείνει μονόπλευρη, χαθήκαμε. Γι' αυτό το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε να φτιάξει τη νέα οδηγία και να την ενδυναμώσει τόσο, διότι οι χώρες μέλη έχουν παραλείψει μέχρι τώρα να αποκαταστήσουν την ισορροπία αυτή και θεωρούν ότι δεσμεύονται μόνο από την θερμή ε, μεταχείριση του επενδυτή. Μόνο αυτόν έχουν υπόψη τους οι Ενώ σε κάθε διάταξη περί εφαρμογής της μελέτης περιβαλλοντικού αντικτύπου υπάρχουν ρητές διατάξεις για τις δαπάνες που θα πρέπει να προβλέπονται, δηλαδή πρέπει να καταθέσει αυτό που ενδέχεται να ρηπάνει το απαραίτητο ποσό για να αποκατασταθεί το περιβάλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μποστινάρο. Δεν ξέρω αν έχει κάτι να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να απαντήσει στις ερωτήσεις. Να παρατηρήσω σε σχέση με αυτό το οποίο είπατε ότι από πλευράς ε, η, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να ελέγξει τα στοιχεία τα οποία αποστέλουν οι Ισπανικές Αρχές και εφόσον δεν επολιθεύονται οι δηλώσεις αυτές και τα στοιχεία υπάρχει η διαδικασία επιπαραλήψη. Και όπως είπα υπάρχει η διαδικασία αποκατάστασης γιατί είναι δεδομένη η υποχρέωση της επιχείρησης να καλύψει την περιοχή και να αποκαθαστήσει ε, την φύση. Πέρα από τα επίσημα στοιχεία λοιπόν τα οποία μας απέστειλαν οι αρμόδιες ισπανικές αρχές ε, σε όλα τα επίπεδα σχετικά με τις απορρίψεις δεν έχουν υπάρξει ε, ίχνη ότι θα καταστεί η περιοχή ε, τουλάχιστον από το διάλογο τον οποίο είχαμε και έχουμε προς τις Ισπανικές Αρχές θα επιμείνουμε γύρω από όλα αυτά τα θέματα. Ε, η αναφέρουσα τελευταία έχει το λόγο. σχετικά με τις πληροφορίες τις οποίες οι διάφορες ε, περιφερειακές ε, υπηρεσίες Έχουμε επίσης και ένα έγγραφο από την Υπηρεσία Ιδάτων της Ανδαλουσίας, το οποίο λέγει ότι η προέλευση των υδάτων στην περιοχή είναι από τις βροχές και όταν πραγματικά παίρνουμε τέτοια στοιχεία στην ε, διάθεσή μας ε, κατανοούμε ότι στην Ισπανία δεν ζούμε σε ένα πραγματικό κράτος δικαίου. Son un problema. Tenemos que ser los ciudadanos, voluntarios y colectivos quienes tengamos que ejecutar el tema que se aplique o bien la directiva Hábitat y demás. Y que eh, otra cosa es que no, o sea, no nos tenemos que tirar ni, ni, por, ni por... Σε σχέση με την Natura 2000 το θέμα είναι ότι έχει δημιουργηθεί ε, και νομολογία η οποία καλύπτει ακριβώς τις ρυθμίσεις ε, για ε, τους υδάτινους πόρους εφόσον θεωρούνται κοινοί υδάτινοι πόροι, κοινή ωφέλειας αν θέλετε η κατανάλωσης και οι οποίοι στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να έχουν βλαφθεί. και υπάρχει χρήση των συγκεκριμένων αυτών υδάτων. Υπάρχει συγκεκριμένη οδηγία για το διαχείριση των υδάτινων πόρων. Ξέρουμε ότι υπάρχει και αντίστοιχη νομολογία και σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο κτλ. Και δεν πρέπει να περιοριστούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα στοιχεία τα οποία παίρνουν από τις Ισπανικές Αρχές. Λοιπόν, θα ήθελα να πω εδώ ότι η άποψή σας είναι σεβαστή, ε, αλλά δεν θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά ότι η Ισπανία δεν είναι ένα κράτος δικαίου, είναι ένα κράτος το οποίο δεν γίνεται σεβαστό το δίκαιο. Κοιτάξτε, αν κάποιος έρχεται εδώ και λέει τέτοια πράγματα, είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να δεχτούμε εμείς στη συζήτηση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ισπανία είναι κράτος δικαίου ε, και δεν πρέπει να λέγονται τέτοια πράγματα. Όπως είπαν και οι άλλοι ομιλητές, θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η, η αναφορά σύμφωνα με τους κανόνες της Επιτροπής μας. Οι πληροφορίες που έχουμε και από την Δημοτική Αρχή του Αλχεσίρας και από την τοπική κυβέρνηση της ε, ε, Ανδαλουσίας έχουν αποσταλεί τέτοια στοιχεία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν θα πρέπει να μας ενημερώσει και μας είχε πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να τεθεί στο αρχείο το θέμα αυτό εφόσον συνεχίζεται η διαδικασία αποκατάστασης της ε, περιοχής. Πάντως νομίζω ότι έχει προχωρήσει η διαδικασία εφόσον υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας τις μεταφέρει και οι πληροφορίες από την τοπική κυβέρνηση και οι πληροφορίες από τις δημοτικές αρχές και ε, θα ασχοληθούμε εκ νέου με το θέμα αυτό με τις πληροφορίες οι οποίες θα προσθεθούν. Εντάξει. Κοιτάξτε, ζητήσατε το λόγο, αλλά ε, πάρα πολύ σύντομα. Προσωπική μου άποψη υπάρχουν δύο θέματα που είναι ενδιαφέροντα εδώ. Το θέμα της αποκατάστασης έχει μεγάλη σημασία. Και θα ήθελα επίσης ε, να ελεγχθεί η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε μέχρι τώρα σε ποιο βαθμό ήταν ε, πράγματι Αυτά θα περιλαμβάνονται στα στοιχεία τα οποία έχει παραλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περνάμε στο επόμενο θέμα τώρα της ημερησίας διάταξης. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα με ενημέρωση για την αποστολή, τη διερευνητική επίσκεψη στην Ελλάδα. Μαλτίνη Παλιαδέλη, Χουντής φαντάζομαι. Έχουν προετοιμάσει ένα έγγραφο. Είναι στα αγγλικά το έγγραφο αυτό, είναι αρκετά μεγάλο. Ξέρετε ότι σε πολύ λίγη ώρα θα πρέπει να συγκαλέσουμε τους συντονιστές και έχουμε και άλλες αναφορές στην παρουσία των αναφερομένων. Το έγγραφο αυτό στην εισαγωγή παρουσιάζει τις διάφορες αναφορές. Para visitar Grecia y που οδήγησαν εν πάση περιπτώσει στο να πάμε στην Ελλάδα και να δούμε επιτόπου ποια είναι η κατάσταση σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται σε σχέση με τις χωματερές βασικά σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας αναφέρεστε στο έγγραφο στο πώς, ε, πότε κατατέθηκαν οι διάφορες αναφορές και υπάρχουν, ε, εναλλακτικές, υπάρχουν ε, αναφορές και στις περιοχές τις οποίες ε, εμείς η αντιπροσωπεία δηλαδή επισκέφθηκε στο ελληνικό έδαφος. Πήγαμε στο γραμματικό στην Αθήνα όπου είχαμε την δυνατότητα να μιλήσουμε και με τις εθνικές αρχές. Συναντήσαμε και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και ζητήσαμε την άποψή του για το τι ακριβώς συμβαίνει. Είχαμε την δυνατότητα να συζητήσουμε επίσης και με τις περιφερειακές αρχές και με τις τοπικές αρχές. Πήγαμε στη μικρή πόλη του Μαραθώνα. Είχαμε την δυνατότητα εκεί να συναντηθούμε με τις δημοτικές αρχές και να επισκεφθούμε τοπικά αυτό το βουνό αν θέλετε στο οποίο είχαν επιστήσει την προσοχή μας ε, οι αναφέροντες ε, τα προβλήματα γενικά τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Θα ήθελα να θυμίσω εδώ ότι την επομένη μέρα πήγαμε στην Πελοπόννησο στη Μεγαλόπολη, συναντηθήκαμε με τον δήμαρχο της Τρίπολης, ήρθαμε σε επαφή ε, και με τους ε, αναφέροντες ε, και στη συγκεκριμένη εγκατάσταση στην οποία υπάρχουν τα προβλήματα. Opinión los peticionarios y con las eh, Είδαμε ποια ήταν η κατάσταση Στην Αθήνα πάλι επισκεφθήκαμε τη Φιλή, πολύ κοντά στην Αθήνα, όπου μαζεύονται, απορρίπτονται γενικά όλα τα απόβλητα της Αθήνας. Και εκεί είδαμε ακριβώς τι σημαίνει και την τρίτη μέρα όπως θα δει κανείς στο κείμενο. Πήγαμε στην Κέρκυρα. Επισκεφθήκαμε τις χωματερές της περιοχές αυτές και μετά πήγαμε στο Καρβουνάρι και στη Λευκήμη με πλοίο. Συναντηθήκαμε με τις τοπικές αρχές Εκεί ήταν και οι τοπικοί δήμαρχοι και μας συνόδευσαν στις χωματερές που υπήρχαν στις ορεινές περιοχές και μας εξήγησαν τα προβλήματα τα οποία είχαν με τις χωματερές αυτές και περιλαμβάνονται όλα αυτά λεπτομερώς στο έγγραφο αυτό και ευχαριστώ εδώ και τη γραμματεία για την προσπάθεια που έκανε για να ε, διανεμηθεί εγκαίρως. Στο τέλος υπάρχουν ορισμένα συμπεράσματα στα οποία καταλήγεται και στο τέλος καταλήγουμε σε συγκεκριμένες συστάσεις με τις οποίες θα κλείσουν οι συζητήσεις τις οποίες θα κάνουμε γύρω από το θέμα αυτό. Δεν ξέρω αν ο κύριος Μαλτίνη μπορεί να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τα στοιχεία θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Μπαλντίνη. Έχετε το λόγο. Έχω... Δεν ξέρω σε ποια γλώσσα να μιλήσω, αγγλικά, κροατικά ή ιταλικά. Θα μιλήσει ακροατικά ο μιλητής. Ήδη ε, Είχα ήδη αναφερθεί ε, σε αυτή την αποστολή που οργανώθηκε στην Ελλάδα. Πρέπει να πω ότι ε, θα ήθελα ειλικρινώς να ευχαριστήσω τον ε, επικεφαλής αυτής της αποστολής, γιατί ηγήθηκε της αποστολής με παραδειγματικό τρόπο. Είχαμε όντως την δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή και με τους αναφέροντες, αλλά και με τις αρμόδιες αρχές. Για να μην μακρηγορήσω και να μην χάσουμε πολύ χρόνο, θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή μου σε μία σύσταση και σε μία πρόταση πρόταση τροπολογίας που σχετίζονται με αυτήν την εξαίρετη εργασία που έλαβε χώρα στην Ελλάδα. Εργασία, λοιπόν, συγγνώμη, πρόταση ε, στην οποία υπογραμμίζω την ανάγκη να αντιμετωπιστεί ε, ε, αποτελεσματικά το, το θέμα των χωματερών στην Ελλάδα. Η κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πρόκειται ε, για ε, ε, αμίαντο που βρίσκεται πλέον σε ασβεστολιθικά εδάφη γνωρίζετε ότι πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό ε, ε, ε, μόρφωμα της Μεσογείου που δημιουργεί σημαντικά προβλήματα όσον αφορά την απορροφητικότητά του στο δημόσιο, στον υδροφόρο συγγνώμη, ορίζοντα. Πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να υπάρξει ευρωπαϊκή βοήθεια έτσι ώστε να διευθετηθεί το ζήτημα διότι είναι πλέον εξαιρετικά επίγον. Σε αυτήν την περιοχή προκύπτει μεγάλος κίνδυνος, κυρίως από τον αμίαντο. Και θα ήθελα να ζητήσω επίγοντα έλεγχο και ταυτόχρονα βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις τοπικές αρχές. ούτως ώστε να λυθεί το συντομότερο δυνατό ε, αυτό το πρόβλημα και να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση η οποία μπορεί να ε, έχει εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις ε, στους γειτονικούς πληθυσμούς. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τους συμμετέχοντες στην αποστολή αλλά και στις ελληνικές αρχές. Θα δώσουμε το λόγο, λέει ο Πρόεδρος, σε διάφορους συναδέλφους. Πολύ γρήγορα, γιατί επίκειται και η συνάντηση των, ε, συντονιστών και έχουμε μετά και μία άλλη αίτηση, ο κύριος Χουντής. Ε, Ωραία, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βέβαια ο χρόνος είναι σύντομος, ε, αλλά θα ήθελα να πω ορισμένες εισαγωγικές παρατηρήσεις και κάποιες αναφορές επί του κειμένου που δουλεύουμε για να δούμε πού θα καταλήξουμε ως Επιτροπή μετέχοντας σε αυτή την Επιτροπή οφίτσιο. Το πρώτο αγαπητοί συνάδελφοι το γράφει το κείμενο, το ανέφερε και ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας. Η επίσκεψη άξιζε τον κόπο. Διότι είδαμε τα σημεία όπου υπάρχουν τα προβλήματα σύμφωνα με τους αναφέροντες. Είδαμε και τη φυλή που ήταν εκτός των αναφορών και βεβαίως από εκεί μπορεί να βγάλει κανείς γενικά συμπεράσματα στο πώς γίνεται η διαχείριση των αποβλήτων. Προσθέτω, επειδή σε αρκετές περιπτώσεις δεν γνώριζαν αυτή τη διαδικασία, ξέρω αγαπητοί συνάδελφοι ότι θα έρθει ένας δεύτερος κύκλος αναφορών από παρόμοιες καταστάσεις στην Επιτροπή μας, διότι αυτό έδειξε έναν δρόμο. Δεύτερη παρατήρηση. Αναφέρεται στην έκθεση και είναι σωστό και γι' αυτό πρέπει να δουλέψουμε με ευθύνη ότι ο κόσμος, οι φορείς, οι αναφέροντες εκεί που επισκεφθήκαμε μας είδαν σαν μια ελπίδα, σαν μια σωτηρία ότι μπορούν να βρουν το δίκαιο τους. Και έτσι είναι. Με τον τρόπο τους, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Το τρίτο, για να είμαι σύντομος, επειδή παρουσιάζεται ως γενικό χαρακτηριστικό στις περιοχές και που έχει να κάνει με τα ρέματα και τον υδροφόρο ορίζοντα όπου το εμφανίζεται στις περισσότερες των περιπτώσεων. Θέλω να σας πω αγαπητοί συνάδελφοι ότι με βάση τραγικά γεγονότα της προηγούμενης εβδομάδας στο νησί της Ρόδου δηλαδή μετά από βροχόπτωση επειδή έχουν μπαζωθεί ρέματα και ποτάμια ξεχύλισε το ποτάμι είχαμε τρία θύματα, τρεις νεκρούς καταστροφές στις περιουσίες. Το συμπέρασμα που θέλω να σας πω αναφέροντας αυτό το τραγικό γεγονός είναι ότι αυτά τα θέματα στην Ελλάδα μπαζώματα, κρύβουμε τα ρέματα. Το πρόβλημα του υδροφόρου ορίζοντα είναι πρόβλημα ζωής ή θανάτου όπως αποδεικνύουν και τα τελευταία γεγονότα. Και επομένως όπου το διαπιστώνουμε στις αναφορές θα έλεγα ότι θέλει μια μεγαλύτερη ευαισθησία στο κατά πόσον γίνονται οι απαραίτητες μελέτες. Τέταρτη παρατήρηση. Κατά τη γνώμη μου, από αυτά που είδαμε και από την τεκμηρίωση προκύπτουν πρώτο ότι οι μεν αρχές δεν μας λένε την αλήθεια έτσι στο κείμενο δεν θα βιαζόμουν να πω ότι έχουν γίνει όπως ισχυρίστηκαν οι αρχές βήματα το τελευταίο διάστημα και θα σας αναφέρω χαρακτηριστικό παράδειγμα δηλαδή υπήρχε μια καθυστέρηση υπήρχαν κομματερές τώρα με στη βιασύνη πρέπει να λύσουμε ορισμένα προβλήματα. έχουμε αρχίσει την ανακύκλωση. Μένω στο τελευταίο και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία διότι ανακύκλωση στην Ελλάδα και με βάση τα στοιχεία που έστειλαν οι αρχές δεν γίνεται. Όποιος τα ακούσει από τους Έλληνες πολίτες θα γελάσει. Μόνο ένα θέμα και εδώ προκύπτει η ευθύνη και της Κομισιόν και δεν ξέρω αν είναι εκπρόσωπος της Κομισιόν και για αυτό το θέμα να απαντήσει αν έχει κινηθεί και έχει κινηθεί σε βάρος της Ελλάδας σύμφωνα με τη διαδικασία pilot πρόβλημα στο κατά πόσον γίνεται σωστά η διαλογή στην πηγή το περίφημο θέμα των μπλε κάδων δεν υπάρχουν τέσσερις κάδοι υπάρχουν μπλε κάδοι ένας κάδος αν αυτό γίνεται σωστά. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι έχει κινηθεί διαδικασία από την πλευρά της Κομισιόν και θα ήθελα να το, θέσει. Πράγμα που βάζει υπό αμφισβήτηση τον ισχυρισμό των αρχών ότι, εν πάση περιπτώσει, έχουμε προχωρήσει και στην ανακύκλωση, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο. Και είναι πάρα πολύ κρίσιμο κατά τη δική μου άποψη. Από εκεί και πέρα θέλω να αναφερθώ, ναι, θέλω να αναφερθώ στην υπόθεση του γραμματικού και πού είναι οι ενστάσεις στο κείμενο. Στο κείμενο που ειναι οι ενστάσει στο κειμενο στο κειμενο που γραφτηκε η μία μου έσταση, ήδη την ανέφερα, είναι η ανακύκλωση. Επιφυλάσσομαι να σας δώσω και περισσότερα στοιχεία ότι δεν στέκει ο ισχυρισμό των ελληνικών αρχών. Ότι δεν γίνεται ανακύκλωση, και το έγγραφο της Κομισιόν το οποίο μπορεί να μας το προσκομίσει ότι πράγματι έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι σχετικά με το γραμματικό, τα λέω επιγραμματικά. Υπάρχει κενό στη δική μας την έκθεση, κενό που δεν έχει απαντηθεί από τις ελληνικές αρχές, ή να το πω καλύτερα από τις συζητήσεις που ακούσαμε η απάντηση επιβεβαιώνει αυτό που ισχυρίζονται οι αναφέρονται στην περίπτωση του γραμματικού ότι κατά την αναθεώρηση της αδειοδότησης δεν ελήφθη υπόψη η αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο της κοινότητας. Δεν τα έχουν πάρει υπόψη. Το ομολόγησαν και αυτό πρέπει να γραφτεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι έτσι όπως τοποθετείτε το θέμα θεωρείτε ότι εντάξει το κάναμε, είχαμε μια αρχική αδειοδότηση ενώ η ένσταση που γίνεται είναι ότι δεν ελήφθησαν υπόψη και μάλιστα κατά αναδρομικό τρόπο όπως περιλαμβάνει η οδηγία του 2008 κάθετος 1 η οποία έπρεπε να είχε ληφθεί και αυτό ισχύει και σε άλλες περιπτώσεις. Το δεύτερο και το λέω πολύ απλά δεν απαντήθηκε το ερώτημα αν στο γραμματικό έγιναν γεωτρήσεις αυτές που έγιναν δεν ήταν στο, από την αρχή της μελέτης στη συνέχεια δεν ήταν στο καταλληλότερο σημείο οι υδρογεωλογικές μελέτες που έγιναν και στηρίχτηκαν από τους καθηγητές οι καθηγητές δεν ήρθαν κατά την ακρόαση να μας υποστηρίξουν αυτή την πρόταση επομένως είναι έολες, έολοι οι ισχυρισμοί ρέματα υπάρχουν όπως το παραδέχονται οι αρχές στην αρχή η περιφέρεια στη συνέχεια είναι η θεωρία η τραγική που είπα καλύπτονται και μετά τα μπαζώνουμε και μετά βλέπουμε τις συνέπειες επομένως εδώ υπάρχουν προβλήματα και τελειώνω, τελειώνω γιατί πράγματι θα μιλήσουν και άλλοι σε μια ακόμα χαρακτηριστική περίπτωση και δεν συμφωνώ πέρα από το καρβουνάρι κτλ. θα αναφερθούν ίσω άλλοι, είναι η περίπτωση τη Λευκήμη. Στη Λευκήμη, αγαπητοί συνάδελφοι, όσοι είμαστε εκεί, όταν είδαμε το κύτταρο, είχε μέσα νερό. Ήταν μια μικρή λίμνη. Έτσι δεν είναι, μια μικρή λίμνη. Ο ισχυρισμό ότι αυτό είναι από τη βροχή δεν στέκει με τίποτα. Δεν στέκει με τίποτα. Αλλά για κάποιον που δεν είναι πιστικό, δεν έχει πιστεί, θα καταθέσω σχετική μελέτη του ΙΓΜΕ που λέει ότι έχουμε υδροφόρο ορίζοντα πολύ ψηλά. Επομένως δεν είχαμε να κάνουμε νερά της βροχής, είχαμε να κάνουμε με υδροφόρο ορίζοντα που επιβεβαιώνει ότι υπάρχει. Γι' αυτό επέμενα και τελειώνω με αυτό ότι αυτό το πρόβλημα με τον υδροφόρο ορίζοντα, με τις γεωτρήσεις που πρέπει να φτάσουν σε βάθος για να το αποκαλύψουν, είναι μία από, τα, μία από τις βασικές, τα βασικά προβλήματα που εμφανίζουν οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην Ελλάδα. Γι' αυτό έχουμε αυτή την πληθώρα των περιπτώσεων εκτός από άλλες ε, περιπτώσεις. Επομένως, οι συστάσεις μας πρέπει να είναι αυτά τα παράνομα έργα πρέπει να δούμε αν θα μπορούν να συνεχιστούν, δεν μπορούν να συνεχιστούν. Ο ισχυρισμό ότι ξοδεύτηκαν χρήματα και τι θα κάνουμε τώρα δεν στέκει, γιατί ξοδεύτηκαν χρήματα και στην περίπτωση τη Σάμου και μετά καταστράφηκαν και πήγε στράφη όλο αυτό το πράγμα. Και δεύτερο, σε ορισμένες περιπτώσεις τουλάχιστον ας γίνουν γεωτρήσεις έτσι όπως πρέπει στο, γραμματικό να αποδειχθούν οι ισχυρισμοί των αναφερόντων και σε άλλες περιπτώσεις και οι συστάσεις πρέπει να είναι ανάλογες από τη δική μας πλευρά. Σταματώ εδώ γιατί ο χρόνος μας είναι περιορισμένος και ε, θα μιλήσουν και άλλοι, ε, βλέπω και τους αναφέροντες και περιμένω και τις απαντήσεις από την Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ε, vamos a ver, vamos έχει ζητήσει και η κυρία Άουκεν το λόγο, πάρα πολύ σύντομα. Ο κύριος Σαγκουράκης, η κυρία Άουκεν και θα πρέπει να δώσουμε το λόγο και σε δύο α, αναφέροντες οι οποίοι περιμένουν. Μέχρι τις 6.30 έχουμε διερμηνία, σας το θυμίζω, το λέω για τους συντονιστές, για τον κύριο Τσίτσεστερ, την κυρία Βέρτμαν, τον κύριο Μποστινάρο. Μήπως θέλετε να το κάνουμε αύριο το πρωί την συνάντηση των συντονιστών. Όχι. Να τελειώσουμε ό,τι ώρα τελειώσουμε τότε χωρίς διερμηνία. Μία φράση λέει η κυρία Οκεν, σύντομα, εξ ονόματος του Χέφνερ, ο οποίος λόγω προβλημάτων μεταφορών δεν μπορεί να είναι μαζί μας. Ήθελε να είναι εδώ, είναι ικανοποιημένος από την παρουσίαση, από την έκθεση. Ε, thank you, ε, Ο κύριος Αγγουράκης έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θεωρώ ότι ήταν μια σημαντική ε, πρωτοβουλία αυτή. Ε, νομίζω όσοι συμμετείχαν στην αντιπροσωπεία είδαν άμεσα πόσο μεγάλα και πόσο σοβαρά είναι τα προβλήματα που σχετίζονται με διάφορες πλευρές του, του περιβάλλοντος. Υπάρχουν πραγματικά και άλλες πολλές περιπτώσεις παρόμοιες ενδεχομένως και πιο σοβαρές ακόμα, αναφέρουμε στην εξόριξη χρυσού παραδείγματος χάρη στην περιοχή των Σκουριών και άλλα σημεία της χώρας και εγώ πιστεύω ότι πράγματι στο μέλλον θα έχουμε και άλλες ε, αιτήσει για ε, επισκέψεις ε, και παρέμβαση. Θεωρώ και εγώ ότι οι ελληνικές αρχές δεν λένε την αλήθεια ή τουλάχιστον δεν λένε όλη την αλήθεια για τα ζητήματα που έθεσε η αντιπροσωπεία ε, στην ε, επίσκεψή της στην Ελλάδα. Ως ε, χαρακτηριστικό παράδειγμα θα αναφερθώ στο παράδειγμα της Ερμιονίδας και της Αργολίδας που βέβαια δυστυχώς η αντιπροσωπεία δεν μπόρεσε να επισκεφτεί η ίδια. Είναι σωστή η περιγραφή που κάνει και ευχαριστώ γι' αυτό. Πράγματι η έκθεση αντανακλά τα πολύ σοβαρά προβλήματα που έχει αυτή η περιοχή Πιστεύω όμως ότι πρέπει η Επιτροπή μας να επιμένει στις αρμόδιες αρχές να τοποθετηθούν στα ζητήματα στα οποία γίνεται η αναφορά, Το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και πρέπει να σας πω ότι ορισμένα από αυτά έχουν επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο όσον αφορά παραδείγματο χάρη το απαράδεκτο, η απαράδεκτη κατάσταση με τα 40.000 ε, πακέτα σκουπιδιών που ε, απλά σκεπάστηκαν με χώματα ε, οξύνοντας ακόμα περισσότερο ε, το πρόβλημα. Κατά συνέπεια νομίζω ότι πρέπει ε, να επανέλθουμε και κλείνοντας θα ήθελα να σημειώσω στα συμπεράσματα στα οποία αναφέρεται η έκθεση ορισμένα είναι σωστά αλλά πιστέψτε μου, το κυριότερο πρόβλημα που υπάρχει στην Ελλάδα δεν είναι θέμα έλλειψης αλληλεγγύης όπως σημειώνεται σε κάποιο σημείο. Αυτό που υπάρχει και σημειώνεται και στην έκθεση, αλλά πρέπει να τονιστεί ακόμα περισσότερο, είναι η βαθύτατη δυσπιστία ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων ε, των εργαζομένων ότι με αυτές τις πολιτικές μπορούν ε, να λυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Έχει όλο και περισσότερο διαδίδεται η άποψη ότι μια ανάπτυξη που εξυπηρετεί το κέρδος, μια άναρχη ανάπτυξη για αυτή που υπάρχει στην Ελλάδα και που υπάρχει και σε άλλες ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα πολύ σοβαρά προβλήματα του περιβάλλοντος και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται, χρειάζεται και πολύ πιο στοχευμένες παρεμβάσεις, χρειάζεται πολύ πιο στενή παρακολούθηση των εξελίξεων και το τι ισχύει και το τι εφαρμόζεται και πολύ περισσότερο χρειάζεται μια πολύ μεγαλύτερη παρέμβαση ε, του λαϊκού παράγοντα ώστε πραγματικά να υπάρχουν τέτοιες λύσεις που να εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να προσθέσω ένα πράγμα. Προφανώς κάνουμε μια προσπάθεια, δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε όλο τον κόσμο. Πραγματικά η προσπάθεια ήταν τεράστια αυτή την οποία κάναμε. Πήγαμε όπου μπορούμε να πάμε, ε, πήγαμε. Ξέρουμε ότι υπάρχουν περισσότερα προβλήματα, ξέρουμε ότι υπάρχουν περισσότερες περιοχές που θα έπρεπε να επισκεφθούμε αλλά η προσπάθεια την οποία κάναμε πράγματι ήταν τεράστια όπως γνωρίζουν οι συνάδελφοι. Κάνουμε προσπάθειες που ίσως άλλες χώρες δεν τις κάναμε. Ο κύριος Γλίκας και ο κύριος Παπαδόπουλος. Ο κύριος Παπαδόπουλος έχει πρώτο το λόγο. Ε, αξιότιμα μέλη, αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές και κυρίες Ευρωβουλευτές, θέλω εκ μέρους όλων των ανθρώπων στην περιοχή της Υπήρου και της Κέρκυρας που επισκεφθήκατε να σας ευχαριστήσω για την φοβερή φοβερή δουλειά και επίσκεψη και το λέω με συγκίνηση που έκανε η Επιτροπή σας. Στην παραμυθιά, σε, ένα, σε, αυτά τα μέρη της Υπήρου, ποτέ, ποτέ μια κοινοβουλευτική επιτροπή τόσο μεγάλη δεν είχε έρθει να αγγίξει τον πολίτη από τόσο κοντά. Σας ευχαριστώ εγώ εκ μέρους όλων αυτών των ανθρώπων για αυτή τη δουλειά σας. Η Επιτροπή Αναφορών είναι πράγματι κοντά στον πολίτη αλλά αναρωτηθήκατε ποτέ εδώ μέσα σε αυτή την Επιτροπή Αναφορών γιατί οι δυο πολίτες που αναφέρουν τα θέματα αυτά στην Ελλάδα είμαι ο κύριος Γκίκας και εγώ που είμαστε μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί. Το γιατί είναι γιατί εγώ και ο Κυριάκος ο Γκίκας δεν έχουμε καμία πελατειακή σχέση με το ελληνικό κράτος και γιατί μακριά από την πατρίδα μας δεν μπορέσαν να μας απειλήσουν με εξοντοτικές μηνύσεις ή επαναλαμβόμενους φορολογικούς ελέγχους. Αυτό είναι μια μικρή παρένθεση. Έρχομαι στο «never in my backyard», γιατί αυτό ακούγαμε συνέχεια από τις ελληνικές αρχές. Κανείς δεν θέλει τα σκουπίδια στην αυλή του. Αυτό είναι ένα άλοθη. Το κανείς δεν τα θέλει στην αυλή του είναι η πιο εύκολη δικαιολογία για να μην προχωρήσουμε σε λεπτομερής αξιολόγηση των δεδομένων και ο κύριος Χουντής αναφέρθηκε στην βασικότερη μελέτη που έχουμε στα χέρια μας για τη Λευκίνη παραδείγματος χάρη, τη μελέτη του ΙΓΜΕ, που δεν αξιολογήθηκε ποτέ ούτε από το ελληνικό κράτος, ούτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θέλω εδώ να καταλάβουν ο κόσμος, όταν λέμε Επιτροπή, λέω Κομισιόν, για να μην μπερδεύουμε τις Επιτροπές. Δεν ήρθαμε γιατί δεν θέλαμε τα σκουπίδια στην αυλή μας Ήρθαμε όταν καταλάβαμε ότι βεβιασμένες διαδικασίες των ελληνικών αρχών για τη χωροθέτηση το χιτά γινότανε μόνο και μόνο με πολιτικά κριτήρια. Ο κύριος Μανιάτης, ο Υπουργός, μας κατηγορούσε γι' αυτό. Εγώ θέλω να ρωτήσω τις ελληνικές αρχές να μου δώσουν ένα όνομα. Ένα όνομα ενός Έλληνα πολιτικού, ενός Έλληνα βουλευτή που έχει το χιτά 130 μέτρα από τα όρια του οικισμού του και που το δέχτηκε και λέει ότι δεν αντιδρούσαμε στις χωματερές, στους ανεξέλεγκτους χώρους. Εμείς δεν αντιδρούσαμε γιατί γνωρίζαμε ότι υπήρχαν τρέχοντες διαδικασίες των ευρωπαϊκών οργάνων και ελπίζαμε επιτέλους ότι θα λήξει αυτό το θέμα διαχείρισης των απορριμμάτων με αυτούς τους νέους σχεδιασμούς. Κάναμε λάθος. Και όμως ήρθαμε πριν γίνουν τα έργα για να προλάβουμε τη ζημιά το 2008 βασίζοντας την επιχειρηματολογία μας στην αρχή της πρόληψης, le principe de précaution. Μάλιστα, όταν στηριχτήκαμε πάνω στην αρχή αυτή, που είναι προήμιο των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Κομισιόν την απέρριψε λέγοντας «Ας γίνει το έργο, ας γίνει η ρήπανση και μετά ελάτε να τα πούμε πάλι, αλλά αφήστε να γίνει η ρήπανση πρώτα». παραβίαση της αρχής της πρόληψης. Κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτές, δεν ήρθαμε γιατί δεν τα θέλαμε αυτά τα σκουπίδια στην αυλή μας. Σας το λέω ειλικρινά, ήρθαμε με βαθύ το αίσθημα της υπευθυνότητας και του χρέους απέναντι στο όραμα που ονομαζόταν Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ θα θέλω να μου επιτρέψετε τρεις μικρές εικόνες και θα είναι πολύ σύντομες, γιατί ειδικότερα στην Ήπειρο στην Ήπειρο, την Ευρώπη τη χτίσαμε με το αίμα μας. Στην παραμυθιά αυτοί οι άνθρωποι τον Ιούνιο του 1944 αποτρέψανε γερμανικές δυνάμεις να ανέβουν στην Ορμανδία με το αίμα μας. Γιατί την Ευρώπη την χτίσαμε με τον υδρότα μας. Αυτός ο άνθρωπος εδώ είναι ο πατέρας μου και αυτό το χτίριο είναι το Μπεγλεμό. Ήρθατε στο Καρβουνάρι, το είδατε. Έχουμε γι' αυτό βαθιά το αίσθημα του χρέους. Γιατί αυτά που είδατε σήμερα στο Καρβουνάρι θα τα βλέπατε αν η Ελλάδα δεν είχε μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι. Αυτά τα παιδιά είναι γεννημένα το 1968, είναι συνομιλικοί μου, είναι εξαδέρφια μου. Αυτή η κατάσταση άλλαξε στην Ήπειρο γιατί υπήρξε η Ευρώπη. Γι' αυτό έχουμε βαθύ αυτό το συνέστημα. Και δεν ήρθαμε απλά γιατί δεν θέλαμε τα σκουπίδια στην αυλή μας ήρθαμε για να υπερασπίσουμε συνειδητά το ευρωπαϊκό όραμα και βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ένα κράτος με ένα κράτος και με μια γενική διεύθυνση περιβάλλοντος της Κομισιόν που μας χλεβάζαν. Τελειώνω. Σε presque fini. Δύο minutes. Που μας... Δύο λεπτάκια ολοκληρώνω. Όταν έστειλα φωτογραφίες στην Κομισιόν μου λέγανε ότι τίποτα δεν αποδεικνύει πως αυτές οι φωτογραφίες είναι από το καρβουνάρι. Μπερδεύαν τον θεσμικό τους ρόλο κάποιοι στην Κομισιόν με τον ρόλο τους σαν υποψήφιοι σε βουλευτικές εθνικές εκλογές. Και αναφέρομαι στον κύριο Χρεμλή. Και ολοκληρώνω με το έργο της Επιτροπής Αναφορών. Τα συμπεράσματα και το πόρισμα που θα βγουν από όλη τη διαδικασία αυτή θα πρέπει πρωτίστως να μην επιτρέψουν σε όσους στηρίχτηκαν στο ψέμα και την απάτη να γιορτάσουν για την αδικία και την ατιμορρησία. Το πόρισμα αυτό πρέπει να αποτρέψει στους χιτά του Καρβουναρίου, της Λευκήμης, του Γραμματικού και όπου αλλού στην Ελλάδα να θαυτεί το ευρωπαϊκό όραμα. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο δημιουργήθηκαν αυτές οι πηγές ρήπανσης δεν μεταλλάσσει μόνο τα απορρίμματα σε στραγίσματα που πέφτουν μέσα ρέματα, αλλά μεταλλάσσει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό σε τέρας και τους πολίτες σε χρυσαυγίτες. Αυτό κύριοι της Κομισιόν είναι το πραγματικό πρόδειλο σφάλμα εκτίμησης. Σας ευχαριστώ. Eh. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γκίκας. Ο κύριος Γκίκας παρακαλώ. Γκίκας. Γκίκας. Ε, Γκίκας. Ε, Very, very shortly, very briefly. Σύντομα σας παρακαλώ αν είναι δυνατόν γιατί δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Yes, yes. Okay. Yeah. Yes, no?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 Ε, ίσως θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε αυτά που θέλετε χωρίς την παρουσίαση σε PowerPoint. Καταρχήν να ευχαριστήσω την Επιτροπή που ήρθατε στην... Ε, που επισκεφθήκατε την Ελλάδα I'm very sorry for the delay. Λυπούμε πολύ για την αργοπορία. Που επισκεφτήκατε που ε, μιλήσαμε στην Αθήνα, μιλήσατε με τους ε, τεχνικούς συμβούλους, μιλήσατε με την Προσινά, με τον κύριο Δημήτρη Δαμάσκο και με τους ε, ανθρώπους που δούλεψαν για όλη αυτή την προσπάθεια. Ερχόμενος εδώ στηρίζω την αναφορά μου, στηρίζω την αναφορά του κυρίου Παπαδογενόπουλου και θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο πράγματα ε, να απαντήσω σε μερικά ερωτήματα όσον αφορά την τελευταία συνεδρία στις 24 Τετάρτου. Ήταν παρόν ε, εκπρόσωποι της Κομισιόν, ήταν εδώ ο κύριος Κρεμλής, ε, ήταν ο κύριος Κουγινιώτης και να αναφερθώ δύο λόγια για το χιτά γραμματικού. Όσον αφορά τις εργοστοσιακές μονάδες στο, στο γραμματικό, στην, συγγνώμη, στην Αττική, που συμπεριλαμβάνει το γραμματικό, την, Γερατέα το, και το Δήμο Φιλής οι τέσσερις εργοστασιακές μονάδες που πρόκειται να κατασκευαστούν είναι δυναμικής 750.000 τόνων. Αυτή τη στιγμή στο λεκανοπέδιο της Αττικής δεν παράγονται περισσότερο από 1.600.000 τόνους. Το ερώτημα είναι ότι όλα τα απορρίμητα, τα ασά, θα καταλήγουν σύμμυκτα και η ανακύκλωση δίνεται σε, είναι στο περιθώριο, δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Όσο αφορά για το γραμματικό, για το έργο αυτό που είδατε και που επισκεφτήκατε, είναι ένα φαραωνικό έργο. Η δυναμικότητά του αρχίσει να σημειωθεί ότι στην Ανατολική Αττική που πρόκειται να γίνει το έργο αυτό, οι κάτοικοι εκεί δεν ξεπερνούν το, τους 200.000 κατοίκους. Σύμφωνα με, τον ευρωπαϊκό μέσον, ε, σύμφωνα με την ε, ευρωπαϊκή στατιστική, ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης δεν παράγει περισσότερα από 500 κιλά. Άρα λοιπόν 200.000 κάτοικοι δεν θα παράγουν περισσότερο από 100.000 τόνους με μηδενική ανακύκλωση. Με απλή εφαρμογή της οδηγίας 98-2008 το σύνολο των απορριμμάτων θα, θα πρέπει να είναι λιγότερα. Στην περίπτωση του γραμματικού που είδατε, και εδώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Χουντή, ότι η ανακύκλωση είναι σε, σε... μηδενική. Πρόκειται να κατασκευαστούν ένα σχητά δυναμικής 127.500 ε, τόνων το, ε, το χρόνο, μια μονάδα βιολογικής ξύρασης 127.500 τόνοι το έτος και ε, ε, ένα, μια μονάδα κομποστοποίησης 40.000 τόνων και ένα κδάι 72.500 τόνοι το χρόνο. Το σύνολο αυτό αγγίζει τους 365.000 τόνους. Δηλαδή περισσότερο από 700 με 750.000 κατοίκου. Και θα ήθελα εδώ να ήταν ο κύριος Κρεμλής, ο κύριος Κινιώτης, να μας πει, εν πάση περιπτώσει, ότι τα, τα έργα αυτά είναι μόνο για την Ανατολική Αττική και δεν θα καταλήγουν απορρίμματα, δεν θα στέλνει απορρίμματα όλη η Αττική. υπάρχει η έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου Σταθμός, 22-2012 για με το ερώτημα αν είναι αποτελεσματική η χρηματοδότηση έργων υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων μέσω διαρθρωτικών μέτρων ω τρόπο βοήθεια προ τα κράτη μέλη ώστε να επιτύχουν τους στόχους της πολιτικής διαχείρισης αποβλήτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία μελέτη η οποία έγινε σε τέσσερα κράτη από Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία και Ρουμανία από 8 περιφέρειες και τα αποτελέσματα δεν ήταν καθόλου ικανοποιητικά. Στην περίπτωση της Ελλάδος έστειλα υπόμνημα, έστειλα επιστολή, ε, έκθεση του κυρίου Δημήτρη Δαμάσκου και μου απαντούν ως εξής. Κύριε Γκίκα, ενδέχεται να υπάρχει σημαντικός κίνδυνος οι τέσσερις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων εφόσον σχεδιαστούν και κατασκευαστούν σύμφωνα με την περιγραφή σας να μην είναι σύμφωνες με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης Πρόκειται για ζήτημα το οποίο έχει ήδη θυγεί από το συνέδριο στην προαναφερθήσα ειδική έκθεση. Θα παρακολουθούμε τη συνέχεια που δίδουν οι υπηρεσίε ε, τη Επιτροπή στι συστάσει τη εν λόγω έκθεση προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη χρήση των πόρων στο μέλλον. yeah. Και ε, έρχομαι, έρχομαι στο γραμματικό. δύο λεπτά. Στην περίπτωση του γραμματικού θα σας δείξω μόνο, έχω προετοιμάσει ένα presentation, δεν θα με φτάσει ο χρόνος, αυτή η φωτογραφία που βλέπετε είναι από τις βροχοπτώσεις του Νοεμβρίου. Αν είχατε έρθει τότε, το, αν τότε το, το Σεπτέμβριο υπήρχαν βροχοπτώσεις, θα βλέπατε αυτές τις καταστροφές. Αυτές είναι βροχοπτώσεις που συνέβηκαν την περίοδο του Νοεμβρίου και η φωτογραφία αυτή εδώ πέρα είναι από χθες. Χθες έβρεξε, υπήρχε μια αρκετή ε, perdón, μεγάλη perdón, perdón, και δείτε τα αποτελέσματα στον ευρωπαϊκό κόλπο. Perdón, se... Συγγνώμη, συγγνώμη κύριε Γκίκα. Oh, No, no, take right. no, put your headphones, please, because I'm going yes, to speak please, in yes. Spanish. Eh, eh, lamento mucho, pero tenemos toda... Εγώ λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά υπάρχουν και άλλοι αναφέροντες που περιμένουν. Έχουμε ξεφύγει πια εδώ και μισή ώρα καθυστέρηση και όπως σας είπα στις μισή σταματούν πλέον και οι υπηρεσίες ε, διερμηνίας μετάφραση κτλ. Αν θέλετε λοιπόν να δώσετε στη γραμματεία τα στοιχεία τα οποία έχετε και η γραμματεία θα μας τα διανύμει στους υπόλοιπους ε, παρόντες βουλευτές. Θα πρέπει να κλείσουμε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη πλέον. Περνάμε στην επόμενη τώρα αναφορά την αναφορά του Μοχάμα Ρεζά Φαρντούμ της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αλληλεγγύη και Δημοκρατία σχετικά με τις περικοπές στην Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση. Δίνω το λόγο στον αναφέροντα. Αγαπητοί συνάδελφοι, η αναφορά αυτή έχει σαν στόχο την διάσωση των θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Δημόσια Υπηρεσία. Ο κύριος Λαμασούρ ανέφερε ότι το Κοινοβούλιο αντιτίθεται στην απόφαση της ε, Προεδρίας, της Φιλανδικής Προεδρίας του 2006 για περικοπές ε, και επομένως ε, δεν έχει συμφωνήσει και με την μετάπτωση των πόρων σε, από τις διοικητικές επιχειρησιακές δαπάνες. Πρέπει να πούμε ότι τα προβλήματα στην Ευρώπη ξεκινούν από εξαιρετικά λίγη ρύθμιση και όχι από την υπερβολική ρύθμιση. Από εκεί απορρέουν τα προβλήματα. στι Βρυξέλλε, περίπου 100.000 θέσει εργασία συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και του διεθνεί ε, οργανισμού. Ε, αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι αν χαθούν 5% των θέσεων εργασία μα, αυτό θα σημαίνει ότι στην ουσία θα χαθούν συνολικά περίπου 5.000 θέσει εργασία στι Βρυξέλλε στο Λουξεμβούργο αρκετές ε, κατηγορίες contract agents ε, ε, πληρώνονται κάτω από τον ελάχιστο εθνικό μισθό ενώ 7.000 Ευρωπαίοι δεν παίρνουν πάνω από 2.000 ευρώ τον μήνα. Υπάρχει μια σκηνή στον Capitalism Love Story του Μουρ που δείχνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά εκατομμύρια εκατομμύρια εκατομμυρίων, τα οποία δεν ξέρουμε πού πηγαίνουν. Ε, ενδεχομένως πηγαίνουν στις χώρες BRIC. Αυτό το εξαγόμενο κεφάλαιο ενδεχομένως ε, θα χρησιμοποιηθεί για νέους εξοπλισμούς ε, ή για εργοστάσια, δεν γνωρίζουμε. Ξέρουμε επίσης ότι είναι πάρα πολλές οι θέσεις εργασίας οι οποίες είναι ανασφάλιστες, είναι ε, μη ασφαλείς. Ε, αντιθέτως, ε, είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι κερδίζουν όλο και περισσότερα χρήματα. Πού πηγαίνουν όλα τα χρήματα αυτά που θα έπρεπε να πηγαίνουν στους εργαζόμενους, με ποιο τρόπο, πού θα πάνε όλοι αυτοί οι περιοδικά εργαζόμενοι όταν θα τελειώσει το συμβόλαιο που έχουν ε, με τα θεσμικά όργανα, πώς είναι δυνατόν ε, να ε, αρνηθούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την ιδιαίτερη γνώση που έχουν λάβει, που έχουν αποκτήσει εργαζόμενοι στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δυνατόν να απαιτήσουμε κάποια στιγμή από τους ανθρώπους αυτούς να δείξουν υπεύθυνη θέση. Είναι γεγονός ότι βεβαίως έχουν αυξηθεί πολύ τα κράτη-μέλη. Αυτή τη στιγμή έχουμε 28 χώρες μέλη. Υπάρχουν όμως χώρες οι οποίες ε, δεν εκπροσωπούνται με αντίστοιχο ε, αριθμό υπαλλήλων όπως άλλες χώρες. Επομένως, ε, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλο έλλειμμα σε αυτή την περίπτωση. Επίσης, έχουμε ιδιαίτερο έλλειμμα στην, στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Φαντάζομαι ότι αυτό θα κάνει να καγχάζουν διάφοροι στην Ουάσιγκτον, στη Μόσχα και σε άλλες πρωτεύουσες. Ε, Βεβαίως υπάρχουν ακόμα κάποια αποθεματικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, για το προσωπικό. Εγώ θα ήθελα ε, να επιστήσω την προσοχή της ε, Επιτροπής σας στον νέο κανονισμό των υπαλλήλων που προτείνει και προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς όμως σωστό προηγούμενο διάλογο με τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των εργαζομένων οι εργασίες, οι διαδικασίες μάλλον γίνονται με ταχύτητα, υποπίεση και σαφώς δεν οδηγούν στο σωστό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ λέει η Πρόεδρος. Ζητεί κάποιος τον λόγο. Ε, εμείς επ' αυτής της δεν ζητήσαμε την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όμως αποφασίσαμε να μεταφέρουμε, να μεταβιβάσουμε μάλλον τα ε, στοιχεία στην Επιτροπή Προϋπολογισμών ως αρμοδία καθήλυν ε, του θέματος. Ε, μας έχουν διαβεβαιώσει ότι ε, σημειώνουν, ελέγχουν προσεκτικά όλα τα σημεία τα οποία ο αναφέρον ανέφερε και τα οποία, στα οποία, για τα οποία μίλησε και έχει ξεκινήσει επομένως μια διαδικασία στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Δεν έχουμε όμως εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μιλήσει για το θέμα αυτό. Θέλει κάποιος το λόγο, αγαπητοί συνάδελφοι, όχι, παραμένει ανοιχτή η αναφορά έτσι ώστε να γίνει η σύγκριση των στοιχείων με την Επιτροπή Προϋπολογισμών και μετά βεβαίως ε, θα ε, συνεχίσουμε τη συζήτηση και θα συνεχίσει και αυτή η αναφορά την πορεία της. Ευχαριστούμε πολύ τον αναφέροντα. Είναι ένα θέμα εξαιρετικά μεγάλη σημασία. Είναι ένα ζήτημα επί του οποίου ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια καλά ισορροπημένη απόφαση η οποία θα αποβεί προς το συμφέρον όλων. Ε, επομένως, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της σήμερα ζητώ από τους συντονιστές να παραμείνουν στην αίθουσα ε, και μόλις ε, ελευθερωθεί η αίθουσα από αυτούς που δεν έχουν δικαίωμα να παραμείνουν ε, θα συνεχίσουμε με τους συντονιστές.